της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης. Χαίρομαι και πάλι να καλωσορίσω τον πρόεδρο Γιούνκερ για την, τον ετήσιο λόγο που μας ε, εκφωνεί για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η στιγμή που κατά τα τελευταία χρόνια είναι σημείο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αναστοχασμό και τον προβληματισμό για το έργο που έγινε πέρσι αλλά και για τα θέματα των καταρχήν κατευθυντήριων γραμμών και των ε, προσανατολισμών για το 2017 που θα συζητηθούν από κοινού και θα καθοριστούν από κοινού. Είναι η δημοκρατική διαδικασία όπως έχει καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα για δεύτερη φορά από εσά κύριε Πρόεδρε θα ακούσουμε τα όσα θα μας πείτε. Είπατε ότι εσείς κύριε Γιούνκερος, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το προϊόν σας το αναφέρω ως παράθεμα είναι το προϊόν μιας διαδικασίας ίασης, μιας διαδικασίας θεραπείας. Ακόμα και αν δεν το θεωρούσαν προϊόν, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 έχετε προαγάγει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και την επιστρέψατε στο σώμα. Είναι μια επιτυχία αυτή αυτής. και ελπίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να πορευθούμε αυτή την πορεία στο μέλλον. Εμείς έχουμε μέσω της ε, τρομερής προσοχής που επικεντρώνεται στα όσα τεκταίνονται στην Ευρωβουλή σήμερα διαπιστώνουμε ότι ο λόγος που θα εκφωνήσετε για την κατάσταση της Ένωσης είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός και στα γεγονότα και στα τεκτενόμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε χωρίς αμφιβολία σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αν όχι σε μια ιστορική καμπή όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία της. Κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, Δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 κρατών ε, στην Βρατισλάβα έχουμε την ευκαιρία ως Ευρωβουλή, αποκοινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσουμε μηνύματα ότι είμαστε ενωμένοι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε επιτακτικά αυτό. Και γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι κατά τις τελευταίες εβδομάδες εργάστηκαν σκληρά για αυτή ε, τον λόγο που θα ακούσουμε. Και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχετε τον λόγο για να μας εκθέσετε την κατάσταση της Ένωσης παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αξιότιμοι συνάδελφοι, πριν από ένα έτος, τον Σεπτέμβριο 2015, στον λόγο για την κατάσταση που εξεφώνησα για την κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσα ότι πολλά ελλείμματα και λήψεις υπάρχουν στην κατάσταση της Ένωσης. Στην Ευρώπη είπα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αρκετή ένωση όπως θα απαιτεί το. Ένα έτος αργότερα <clears throat> ισχύει η ίδια αυτή η διαπίστωση. Παρόλες τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε ανιούσα πορεία. Πολλά δεν τροποποιήθηκαν, δεν αλλάξαν προς το καλύτερο. Και υπάρχει και η υπόθεση ότι βρισκόμαστε σε μια υπαρξιακή κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλαπλά και πολυσχηδώς. Ο αριθμός των τομέων και των πεδίων όπου αυθόρμητα ή και όχι αυθόρμητα συμπίπτουμε είναι υπερβολικά μεγάλος. Ο τομέας των πεδίων όπου με αλληλεγγύη συνεργαζόμαστε είναι πάρα πολύ μικρός. Πέρα από αυτά, σε αποκλειστικά εθνικό, εθνικό συμφέρον δίνεται πάντα η προτεραιότητα προ όφελο του εθνικού συμφέροντος για να μην υπάρξει παρερμηνία. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί βέβαια εις βάρος των κρατών μελών. Όχι. Δεν μπορεί κανείς με τα λοστάρια ή με, ε, δια της βίας να επιβάλλει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να είναι άχρωμη και ανούσια η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, σπονδύλους και προσωπικότητα. Έχει πολυσχηδή χαρακτήρα και πολυμορφία. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον στόχο, ακόμα και αν πολλοί το ισχυρίζονται αυτό, να καταργήσουν να καταργήσει τα εθνικά κράτη ή να επιβάλλει θέσεις. Δεν είμαστε εμείς ε, ε, αυτοί που θα διαλύσουν ή θα καταστρέψουν. Είμαστε επικοδομητικοί. Επικοδομούμε και θέλουμε μια καλύτερη, βελτιωμένη Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται στην πορεία της ε, και η Ευρώπη δεν μπορεί ποτέ να γίνει ένα εθνικό κράτος ή να εξομοιωθεί με ένα τέτοιο κράτος. Και πολλές φορές υπάρχουν ρογμές και προβλήματα. Και πολλές φορές ε, υπάρχουν και ε, φόβοι για το τι μπορεί να συμβεί. Αυτό ανοίγει ε, την πορεία στην καλπάζουσα λαϊκιστική τάση που πρέπει να αναχαιτιστεί. Ο λαϊκισμός δεν επιλύει προβλήματα. Το αντίθετο, ο λαϊκισμός δημιουργεί προβλήματα και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν τον λαϊκισμό. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή που ήρθε να κάνουμε μια τίμια, έντιμη επισκόπηση της κατάστασης. Η ανεργία στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή. Μεταξύ 2013 και σήμερα 8 εκατομμύρια νέα, νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και η απασχόληση είχε ανωδική πορεία. Όμως παρόλα αυτά η κοινωνική αδικία παραμένει στην Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει ταχύτατα να δράσουμε και να ε, δράσουμε στους πυλώνες, ε, θεμελιώδεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενέργεια για παράδειγμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η Ευρώπη δεν είναι αρκετά κοινωνική στο πρόσωπο και στο χαρακτήρα της. Αυτό πρέπει να αλλάξει επιτέλους. Die τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθούν να είναι όσον αφορά τις ελλείψεις υπερβολικά υψηλά. Παρότι τα επίπεδα ελλημάτων από κατά μέσο όρο 6,3% του 2009 έχουν μειωθεί σε 1,9% εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα. Το σύμφωνο σταθερότητας δείχνει ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να γίνει όμως σύμφωνο ελαστικότητας. Πρέπει με ελαστική ευφυΐα, με, με να ε, το χειριζόμαστε το μέσο αυτό όσον αφορά την ευληγησία του, ώστε να μην ε, αποτελεί πρόσκομα, εμπόδιο για την επισκόπηση της Ένωσης πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και σε εκείνους που μας παρατηρούν από μακριά. Οι φίλοι και οι εταίροι μας στην παγκόσμια σκηνή που όλοι εξέφρασαν τη θλίψη τους για το Brexit διαρωτώνται με ανησυχία μήπως η απόφαση αυτή των Βρετανών θα μπορούσε να είναι η απαρχή μιας διαδικασίας ε, διάλυσης ε, της ε, διάβρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω, το σεβόμαστε αλλά και θλιβόμαστε ταυτόχρονα την απόφαση που έλαβαν οι Βρετανοί. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει στην υπόστασή της. Θα χαιρόμασταν βέβαια αν <clears throat> το αίτημα αποχώρησης της Βρετανίας υποβαλόταν το δυνατόν ταχύτερα, ώστε να σταματήσουν οι αβεβαιότητες και οι ανασφάλειες που υφίστανται σήμερα. Και για να μπορέσουμε τη σχέση μας προς τη Μεγάλη Βρετανία να, να εξακολουθήσουμε να τις έχουμε σε ένα φιλικό πλαίσιο πρέπει να τις, να τις αναδιατάξουμε. Σε αυτή την αναδιάταξη ανήκει ότι μόνο εκείνος θα έχει απεριόριστη πρόσβαση στην ενιαία εσωτερική αγορά που αναγνωρίζει και εφαρμόζει την ελευθερία κυκλοφορία των ατόμων. Δεν θα υπάρξει μια αλακάρτα ενιαία εσωτερική αγορά για κανέναν. Οι εταίροι μας μας προσεγγίζουν διαρκώς με το ερώτημα τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχει την προθυμία και την ικανότητα να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Είμαστε η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη παγκόσμια. Έχουμε με 140 χώρες συμφωνίες που έχουμε συνάψει. Δεν είμαστε τυφλός, φανατικός, ε, ε, φανατικό τυφλό ενεργούμενο. Είμαστε υπέρ του ότι η συμφωνία για την ανάπτυξη δεν μπορεί να υπονομεύεται από τις συμφωνίες ε, της εμπορικές και εμπόριο σημαίνει μεγαλύτερη, περισσότερες θέσεις απασχόλησης. 30 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτώνται από τις εξαγωγές μας. Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας από τις εξαγωγές μας σε άλλα μέρη του κόσμου εξαρτώνται. Έχουμε τεράστιο όγκο στις εξαγωγές που δημιουργεί επιπλέον 14.000 θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους, κυρίως για αυτούς τους λόγους είμαι έντονα υπέρ του να ολοκληρωθεί η συμφωνία, η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Είναι η καλύτερη συμφωνία που έχουμε συνάψει ποτέ ως ΕΕ, αυτή με τον Καναδά. Τα εχέγγυα που χρειαζόμαστε στις διαφορετικές φάσεις επικύρωσης μπορούν να αποσαφινιστούν και τα προβλήματα και επιφυλάξει μπορούν να αρθούν. Όμως ε, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια επαναχώρηση όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις με τον Καναδά ή νέες διαπραγματεύσεις. Οι εταίροι μας παγκόσμια, κυρίως στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, αλλά επίσης και στην Ινδία και στην Ιαπωνία, μας ε, κρατούν τον καθρέφτη για την προσπάθεια προστασίας του κλίματος ενώπιον μας μπροστά στο πρόσωπό μας. Πρέπει λοιπόν η Παγκόσμια Συμφωνία να αναγνωρίσουμε ότι χωρί τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε συναντήσει. Ήμασταν εμεί πρωτοπόροι και προπομπή. Και καμιά φορά καλέσαμε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο άλλους να κινητοποιηθούν. Τώρα Αμερικανοί και Κινέζοι κινούνται και τώρα πού βρισκόμαστε εμείς υπάρχει το αίτημα της επικύρωσης. Ζητείτε λοιπόν αυτή η συμφωνία για την προστασία του κλίματος επιτέλους να επικυρωθεί. Κάθε καθυστέρηση στην επικύρωση η ε, οποιαδήποτε εργεία θα μας γελιοποιήσει όσον αφορά τη διεθνή σκηνή. Με τους εταίρους μας έξω και με εκατομμύρια Ευρωπαίους στην ίδια την Ήπειρο που παρακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και που μεταξύ αυτών των διαδικασιών πρέπει να βρουν τις λύσεις. Δεν είμαστε εμείς οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ο λόγος που εκφωνώ εδώ σε σχέση με τον λόγο που εκφωνεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την State of the Union, την κατάσταση των ΗΠΑ της Ένωσης, ε, δεν έχει καμιά σχέση. Είμαστε πολύ πιο πολύμορφοι από τη ΣΥΠΑ εμείς και διαφορετικοί από τη ΣΥΠΑ. Όμως η ιστορία, η δεινή, σκληρή ιστορία της Ευρώπης μας έκανε αυτό που είμαστε σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος τα πράγματα να τα καταστήσουμε ακόμα πιο περίπλοκα και ακόμα πιο δυσνόητα από ό,τι είναι. Και μια, ένας λόγος υπέρ της Ευρώπης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> θα απαιτούσε και θάρρος. Όμως οι λόγοι υπέρ της Ευρώπης πρέπει από όλους να εκφωνούνται στα εθνικά κοινοβούλια με θάρρος. In Brüssel laut Τις ε, Βρυξέλλες ε, με την ε, προσπάθεια σαν να λέει κανείς ότι δεν υπήρξε συμμετοχή στην κοινή λήψη απόφασης. Είναι αυτό το αντίθετο ακριβώς από την συνεκτικότητα και την συνέπεια αν συμβαίνει οι πολίτες της Ευρώπης ε, δεν επιτρέπεται περισσότερο να ε, απατώνται, να πλανώνται. Πρέπει να είμαστε έντιμοι μαζί τους για να τους πούμε την αλήθεια. Σε σχέση με τις ε, θεσμικές τριβές βαρέθηκαν οι πολίτες πια. Δεν θέλουν τις αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών και θεσμικών οργάνων και δεν θέλουν με κανένα τρόπο να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Οι πολίτες αναμένουν από την Ευρώπη χειροπιαστά αποτελέσματα με βάση δίκαιες αρχές και αξίες. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ αυτό το οποίο θέλω να προτείνω είναι κάτι το θετικό. Θέλω συγκεκριμένες ενέργειες για τους επόμενους 12 μήνες. Πιστεύω ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι αποφασιστικός αν θέλουμε να επανεκκινήσουμε την Ένωση, αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, οι οποίες φάνηκαν τους τελευταίους μήνες να ενισχύονται. Πρέπει να το κάνουμε αυτό με αποφασιστικό και γρήγορο τρόπο και σε τομείς που έχουν σημασία και έτσι θα δείξουμε στην παγκόσμια σκηνή ότι είμαστε μια δύναμη ικανή ακόμα και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε περισσότερο. Έστειλα μια τέτοια επιστολή και προς τον πρόεδρο ε, Σούλτς και τον πρωθυπουργό κύριο Φίτσο. Οι επόμενοι 12 μήνες είναι οι κρίσιμοι μήνες για μια καλύτερη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που προστατεύει και διατηρεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Μια Ευρώπη που δίνει εμπιστοσύνη, εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες της και αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής πρέπει να διατηρηθεί. Υπάρχουν ερωτηματικά για το τι σημαίνει να είναι κανένας Ευρωπαίος σήμερα, τι σημαίνει να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την Ένωση των Ευρωπαίων. Καταρχάς πρέπει να θυμόμαστε γιατί ε, οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνεργαστούν. Γιατί ξεκίνησαν τις ε, περαιτέρω προσπάθειες ε, για συνεργασία ε, και με τις χώρες όπως η Πολωνία με την οποία πάντα θέλουμε να συνεργαζόμαστε γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Η σημαία στην Ισπανία, στην Πορτογαλία ποιήθηκε για να καλωσορίσει τις χώρες αυτές στη δημοκρατία και στην ελευθερία. Να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει και στην ένωση, επανένωση της Κύπρου. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ υποστηρίζω τους δύο ηγέτες έτσι ώστε να γίνει και να γίνει τώρα. Η Ευρώπη κυρίως σημαίνει η ειρήνη. Δεν είναι τυχαίο ότι η πιο μακρά περίοδος ειρηνική στην Ευρώπη ξεκινά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 70 χρόνια ειρήνη στην Ευρώπη. Σε έναν κόσμο με 40 ανοιχτές πολεμικές σειράξεις που κάθε χρόνο κοστίζουν τη ζωή σε 200.000 ανθρώπους. Φυσικά έχουμε και πολλές διαφορές μεταξύ μας ε, και ε, αντιμαχόμεθα ο ένας τον άλλο, αλλά το κάνουμε με λέξεις, το κάνουμε μέσω του λόγου και όχι μέσω των χαρακομάτων. Οι αξίες μας είναι η βάση αυτού του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Ελευθερία, κράτος δικαίου, δημοκρατία. Οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούσαν να αποδεχθούν ποτέ οι Πολωνοί εργάτες να διώκονται και πολλές φορές να δολοφονούνται στους δρόμους του Έσεξ. Εμείς οι Ευρωπαίοι λοιπόν είμαστε και κατά της θανατικής ποινής. Πιστεύουμε επίσης σε ανεξάρτητα δικαστικά και αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρώπη προωθεί παντού το κράτος δικαίου. Τα προσωπικά μας δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από ισχυρές νομικές διατάξεις. Δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να παρακολουθούνται οι συνδιαλέξεις τους. Δεν θέλουν οι εταιρείες να παρακολουθούν κάθε κλικ στο ποντίκι του υπολογιστή τους και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή προστασία των δεδομένων. Η ιδιωτικότητα μετράει στην Ευρώπη. Also means... Το να είσαι Ευρωπαίος επίσης σημαίνει το εξής. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο για την ίδια δουλειά στον ίδιο τόπο. And this is why... Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πρόταση για τις ε, μετακινήσεις των εργαζομένων και τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο χώρος όπου οι εργαζόμενοι θα γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης με χαμηλά επίπεδα προστασίας. Δεν είμαστε η άγρια δύση ε, του κοινωνικού ντάμπινγκ. Απαιτείται να υπάρχει λοιπόν μια δίκαιη αντιμετώπιση και για την προστασία των καταναλωτών από τα καρτέλ και τις μεγάλες πανίσχυρες επιχειρήσεις. Και κάθε επιχείρηση, είτε μικρή είτε μεγάλη, θα πρέπει να πληρώνει τους φόρους της εκεί που βγάζει τα κέρδη της. Σας υποσχέθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πολεμήσει την φοροαποφυγή. Πολλοί από εσά δεν με πιστέψατε. Αυτό είναι όμως που προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις μας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Oh. Το να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει να ορθώνεις τον άστημά σου απέναντι στην ε, χαλιβουργία. Έχουμε 37 μέτρα αντι-dumping για να προστατεύσουμε τη χαλιβουργία μας από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, γιατί η υπερπαραγωγή σε ορισμένα μέρη του κόσμου δημιουργεί προβλήματα για τους Ευρωπαίους, κλείνει ευρωπαϊκές εταιρείες και διώχνει τους Ευρωπαίους από τις δουλειές τους. Γι' αυτό ακριβώς πήγα στην Κίνα δύο φορές φέτος, για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα του πλεονάζοντος δυναμικού, της πλεονάζουσας παραγωγής. Γι' αυτό πρότεινε η Κομισιόν να αλλάξουμε τον κανόνα του ελάσσονος ε, δασμού. Θέλουμε όλοι σας να υποστηρίξετε την Κομισιόν και να διατρανώσουμε και να δυναμώσουμε τα αμυντικά μας ε, εργαλεία. Θα πρέπει να απαντήσουμε στο dumping όσο ε, δυναμικά απαντούν και οι Αμερικανοί. Είναι και αυτός ένας από τους τρόπους ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γεωργία, η Κομισιόν είναι στο πλευρό των ακροτών. Στις δύσκολες στιγμές. Στο παρελθόν όπως και σήμερα. Πέρυσι ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετώπισε τα προ... τους φραγμούς της ε, Ρωσίας. Γι' αυτό κινητοποίησαμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ υπέρ των αγροτών για να τους ε, βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Γιατί δεν θέλω το γάλα να είναι φθηνότερο από το νερό. Δεν το δέχομαι αυτό. Το να είσαι Ευρωπαίος, για τους περισσότερους από εμά σημαίνει και ευρώ. Με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το ευρώ μας προστάτευσε από χειρότερη αστάθεια. Το ευρώ είναι από τα μεγάλα παγκόσμια νομίματα και μας φέρνει τεράστια οικονομικά ωφέλη. Γλιτώσαμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ χάρη στην ε, νομισματική πολιτική της ε, ΕΚΤΑ. 50 δισεκατομμύρια που, θα μπορούσαν, που μπορούν οι κυβερνήσεις να επενδύσουν στην οικονομία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους. Και μάλιστα οι πέντε πρόεδροι με την έκθεσή τους για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης περιγράφουν την ε, φιλοδοξία της Κομισιόν, η οποία και την υμνούν. Θα ήθελα όλα αυτά να λέγονται πιο συχνά, παντού στην Ευρώπη. Όταν παίρνουν το λόγο οι πολιτικοί, καλό θα ήταν να τα λένε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει μόνο να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, αλλά να ενισχύσουν να ενισχύσει και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν. Θα πρέπει να φτιάξω μια Ευρώπη με δυνατούς πολίτες και δυνατή οικονομία. Και σήμερα αυτό σημαίνει ψηφιοποίηση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ψηφιακή οικονομία αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής. Θέλουμε απλώς πρόσβαση σε ένα ίντερνετ υψηλής ταχύτητας. Θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι. Η οικονομία μας το χρειάζεται. Ο κόσμος το χρειάζεται. Και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή τη ε, διασύνδεση. Τώρα, γι' αυτό ακριβώς σήμερα η Κομισιόν προτείνει μια μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών τηλεπικοινωνίας. Θέλουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις για τις διασυνδέσεις. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη για τα επόμενα 20 χρόνια. Γιατί αν οι Ευρωπαίοι επενδύσουν σε τέτοια δίκτυα και τέτοιες υπηρεσίες, αυτό σημαίνει την, επόμενη δεκαετία έξτρα ένα εκατομμύριο νέες θέσεις απασχόλησης. Η διασύνδεση θα πρέπει να είναι υποφελής για όλους. Γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει ένα, πληρες πλήρες 5G που θα είναι έτοιμο μέχρι το 2025 έχει το δυναμικό να δημιουργήσει επιπλέον 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένα θα υποφεληθεί από την διασύνδεση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι όπου και να ζει, όσα και να βγάζει έχει σύνδεση. Προτείνουμε λοιπόν κάθε πόλη να έχει τέτοια πρόσβαση στο ασύρματο ίντερνετ μέχρι το 2020. Καθώς η δουλειά γίνεται επίσης ψηφιακή, θα πρέπει και οι δημιουργοί μας και οι καλλιτέχνες μας να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία και να προστατεύσουμε τις δουλειές τους. Γιατί είναι το κόσμημά μας οι καλλιτέχνες. Η δημιουργία περιεχομένου δεν είναι χόμπι, είναι επάγγελμα. Θέλω οι δημοσιογράφοι, οι συγγραφείς να πληρώνονται δίκαια για τη δουλειά που κάνουν. Είτε τη δουλειά την κάνουν στο σαλόνι τους, στο στούντιο, είτε το Είτε δημοσιεύεται το έργο τους στο web, στο δίκτυο δηλαδή, είτε σε βιβλίο. Ακριβώς αγαθούμε για αυτή τη δίκαιη αμοιβή. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας σημαίνει επένδυση όχι μόνο στις διασυνδέσεις, αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα 350 δισεκατομμύρια ε, της ευρώ ε, που συμφωνήσαμε έχουν ε, από αυτά έχουν επωφεληθεί χιλιάδες θες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή την πλατφόρμα θα την πάμε πιο πέρα τώρα. Σήμερα προτείνουμε να διπλασιάσουμε τη διάρκεια του Ταμείου και να διπλωσιάσουμε το δυναμικό του, το, τα λεφτά δηλαδή. Θα εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα δώσει τουλάχιστον 500 ε, δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Και θα κάνουμε και ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για να φτάσουμε τα, 300, τα 630 ε, δισεκατομμύρια μέχρι το 2022. Με τη συνεισφορά των κρατών μελών μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο ακόμα πιο γρήγορα μαζί μας τις προσπάθειες για την, ε, θα προσπαθήσουμε για να ελκύσουμε ε, ιδιωτικέ επενδύσει, πρέπει να φτιάξουμε και το κατάλληλο ε, περιβάλλον. Οι ευρωπαϊκέ τράπεζε δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι δύο χρόνια πριν. Αλλά βελτιώνονται σιγά σιγά χάρη στις κοινέ μα προσπάθειε, γιατί χρειαζόμαστε τι τραπεζέ μα. Η οικονομία μας που εξαρτάται σχεδόν ε, αποκλειστικά από τη σταθερότητα των τραπεζών και τον δανεισμό τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρίσκονται οι τράπεζες αυτές σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν είναι και η ώρα να επιταχύνουμε τη δουλειά μας ε, για την Ένωση των Κεφαλαίων Η Κομισιόν ετοιμάζει έναν οδικό χάρτη και θα σας το υποβάλει σήμερα. Μία τέτοια ένωση Κεφαλαίων αγορών θα καθιστά το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα πολύ πιο ανθεκτικό θα δώσει στις εταιρείε μεγαλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στην πίστη, στην πίστοση. Φανταστείτε ότι είστε νεοφυής επιχείρηση και ότι χρειάζεσαι ε, δάνειο. Και η τράπεζα σου λέει όχι. Τώρα δεν έχει πολλέ άλλε επιλογέ. Με την ένωση αυτή όμω των κεφαλαιογορών θα έχουμε επιλογέ. Θα έχουμε δυνατότητε χρηματοδότηση, ώστε οι νεοφυεί επιχειρήσει να στηθούν στα πόδια του. Ε, θα έχουμε τέτοια χρηματοδότηση ε, ρηψοκίνδυνων ε, οικονομικών εγχειρημάτων. Η πρότασή μας για την τιτλοποίηση έχει υποβληθεί εδώ και ένα χρόνο. Έχει το δυναμικό να δώσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σας παρακαλώ να επιταχύνουμε την υιοθέτηση. Το επενδυτικό σχέδιο είναι το καλύτερο, καλύτερο από ό,τι περίμενε οποιοδήποτε Ευρωπαίος. Και τώρα θα αποκτήσει παγκόσμια διάσταση. Σήμερα ετοιμάζουμε μια φιλόδοξη ε, επενδυτική προσπάθεια για την Αφρική και την γύρω περιοχή που μπορεί να συγκεντρώσει 44, 44 ε, δισεκατομμύρια επενδύσεις. Και μπορεί να φτάσει τα 88 εάν ε, βάλουν και τον οβολό τους τα, τα κράτη-μέλη. Θα αντιμετωπίσουμε έτσι μία από τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης. Αν υπάρξει οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες, ε, θα, βοη, θα τις βοηθήσουμε. Γιατί σήμερα είναι πολύ χαμηλή η ανάπτυξή τους και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι και βάζουν σε εκείνο τη ζωή τους, να μείνουν στις χώρες τους. Αυτό πρέπει να γίνει. As much as we Όσο περισσότερο επενδύουμε στη βελτίωση της ε, εργασίας, θα πρέπει να επενδύσουμε και για να απαντήσουμε στο πρόβλημα της, ε, με την ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει να επενδύσουμε στους νέους μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει η Ήπειρος όπου οι νέοι είναι άνεργοι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι Δεν θα δεχτώ ότι μία ολόκληρη γενιά θα είναι η πρώτη γενιά σε 70 χρόνια που θα είναι πιο φτωχή από τους γονείς της. Φυσικά αυτό είναι κυρίως δουλειά των εθνικών κυβερνήσεων. Και εσείς δεν είστε τμήμα από ό,τι ξέρω. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και τις προσπάθειες των κρατών. Το κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για την Νεότητα που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια η Κομισιόν, ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της ε, εγγύησης. Πάνω από 9 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά ή βρήκαν κάποια μαθητεία ε, ή ξεκίνησαν την κατάρτισή τους χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε σε όλη την Ευρώπη την εγγύηση αυτή κυρίως για τις ε, μαθητείες, που βελτιώνουν τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και φτάνουν σε ανθρώπους ε, νέους που την έχουν ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης μπορεί να συνεισφέρει για να βοηθήσει να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους. Υπάρχουν πολλοί νέοι στην Ευρώπη που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνία και να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η λέξη αλληλεγγύη αναφέρεται 16 φορές στις συνθήκες. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μας είναι η απόδειξη αυτής της αλληλεγγύης. Η Ευρώπη είναι μια έκφραση αλληλεγγύης. Και η αναπτυξιακή μας πολιτική είναι ένα έντονο μήνυμα που δίνει προς τα έξω αλληλεγγύης. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κρίση και με την αλληλεγγύη. Και είμαι πεπισμένος ότι πολύ περισσότερη αλληλεγγύη χρειάζεται. Ξέρω όμως ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι θελοντική. Πρέπει να έρχεται από καρδιάς. Δεν μπορεί να εξαναγκάσεις κάποιον και να επιβάλλεις σε κάποιον την αλληλεγγύη. Κάνω έκκληση στη Σλοβακική Προεδρία να γεφυρώσει τι διαφορέ ανάμεσα σε εκείνου που είναι απρόθυμοι να δεχτούν τους πρόσφυγε στις κοινωνία τους και σε εκείνου που είναι πεπισμένοι όπω εγώ ότι ο καθένα πρέπει να σηκώσει ένα δίκαιο μερίδιο. Ε, και πώ γίνεται αυτό μέσω της ε, εγκατάστασή του, Θέλω μια γρήγορη και άμεση ε, δράση και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα για να ε, προστατεύσουμε τους ασυνόδευτους ανήλικους. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να το κάνει. Αλλιώς προδίδει τις αξίες υπό το ίδιο πνεύμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την δημιουργία Ενό σώματο Ευρωπαϊκή αλληλεγγύης. Οι νέοι της Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν εθελοντικά να βοηθήσουν εκεί όπου απαιτείται περισσότερο για να ανταποκριθούμε σε κρίσεις όπως η μεταναστευτική κρίση ή οι σεισμοί στην Ιταλία σαν παράδειγμα. Θέλω το σώμα αυτό των Ευρωπαίων εθελοντών να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό και θέλω το 2020 να έχει 120.000 μέλη με την εθελοντική του συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα αυτοί οι νέοι θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους, θα αποκτήσουν εμπειρίες και θα ζήσουν μια πραγματικά ασύγκριτη ανθρώπινη εμπειρία. Monsieur... Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω στα γαλλικά. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να προστατεύει και αυτή η Ευρώπη θα μπορεί να αμήνεται και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του εδάφους της. Πρέπει να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας και είναι βασική προτεραιότητά μας απέναντι στην τρομοκρατία. Από το 2004 έχουν υπάρξει 30 τουλάχιστον σημαντικές τρομοκρατικές επιθέσεις, 14 τα τελευταία χρόνια. Εμείς ήμασταν αλληλέγγυοι στο πένθος, αλλά θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και στην συνολική μας κοινή απάντηση. Απέναντι στο χείριστο θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πιστοί στις αξίες μας, στις πολυπίκυλες, ανεκτικές, ανθεκτικές και δημοκρατικές κοινωνίες μας. Οι τρομοκράτες δεν θα έχουν καμία πιθανότητα να πετύχουν απέναντι σε αυτές τις αξίες. Η αξία αυτή της ανοχής, σαν παράδειγμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της ασφάλειάς μας και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρώτη στιγμή υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ασφάλεια. Εμείς προχωρήσαμε σε προτάσεις και για τις ποινικέ ευθύνες και για την επαναπροώθηση των ξένων ε, μαχητών. Πήραμε μέτρα για την χρήση των πυροβόλων όπλων και για, τα, για τη χρηματοδότηση του, της τρομοκρατίας, για τον έλεγχο του διαδικτύου ε, σε επίπεδο τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και καταπολεμούμε επίσης και την ριζοσπαστικοποίηση στα σχολεία και στα σοφρονιστικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Έχουμε πολλή δουλειά όμως να κάνουμε ακόμα. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που περνούν στα σύνορά μας. Γι' αυτό υπερασπιζόμεθα τα σύνορά μας και με τη βοήθεια της νέας υπηρεσίας ακτοφυλακής. Η Frontex έχει 600 άτομα στην Ελλάδα σαν παράδειγμα στα σύνορα με την Τουρκία και 100 στην Βουλγαρία. Θα πρέπει να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα για την δημιουργία και την θέση σε λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Ήδη από τον Οκτώβριο θέλω να έχω 250 νέους σύνοριοφύλακες στα εξωτερικά σύνορα της Βουλγαρίας σε αυτή την περίπτωση. Υπερασπιζόμεθα επίσης και ένα <clears throat> και μια σωστή και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για τον έλεγχο των συνόρων. Κάθε φορά που κάποιος μπαίνει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγαίνει από αυτήν θα καταγράφεται το πότε, το πού και ο λόγος των μετακινήσεών του. Μέχρι τον Νοέμβριο θα προτείνουμε ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης των μετακινήσεων, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα δηλαδή, το οποίο θα καθορίζει το ποιος θα μπορεί να ταξιδεύει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα γνωρίζουμε ποιος έρχεται στην Ευρώπη πριν καν έλθει αυτός ο άνθρωπος στην Ευρώπη. Η ασφάλεια των συνόρων Σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών και την αμοιβαία ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε και τις δικές μας υπηρεσίες όπως επίσης και τις εθνικές υπηρεσίες καταστολής των ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων ενημερώνοντας σωστά. Πρέπει όμως να έχουμε τα μέσα των φιλοδοξιών μας στη διάθεσή μας. Θέλουμε μια Ευρώπη που προστατεύει, θέλουμε μια Ευρώπη που αμήνεται, να προστατεύουμε όμως τα συμφέροντά μας και πέραν των σύνορων μας. Ο κόσμος μεγαλώνει συνεχώς. Η Ευρώπη γίνεται όλο ένα και πιο μικρή καθημερινά και δημογραφικά και οικονομικά. <clears throat> Αν θέλουμε να κρατήσουμε την επιρροή μας στον κόσμο, είναι απαραίτητο ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνο από κοινού. Όμως Ακόμα και αν η Ευρώπη είναι υπερήφανη γιατί είναι μια ήρεμη μεγάλη δύναμη, αυτό δεν αρκεί. Στα πλαίσια μιας παγκόσμιας σκηνής, περίπλοκης και πολλές φορές επικίνδυνη. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Συρία. Οι συνέπειες της Συρίας για την Ευρώπη είναι άμεσες. Πού είναι λοιπόν η Ένωση εκεί. Πού είναι τα κράτη-μέλη της Ένωσης στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση της κατάστασης στη Συρία. Η Φεντερίκα Μογκερίνη, η τη εκπρόσωπος για εξωτερικές υποθέσεις της Επιτροπής και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, κάνει μια εξαιρετική μα εξαιρετική δουλειά. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια πραγματική υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια υπουργός Μια υπουργό έλεγα η οποία συγκεντρώνει και εκπροσωπεί και μιλάω για τη Φεντερίκα, τις δυνάμεις συνολικά των εθνικών διπλωματικών μας υπηρεσιών. Έτσι θα αποκτήσουμε μεγαλύτερο βάρος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Συρία θα πρέπει η Φεντερίκα να έχει θέση ε, στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Συρίας. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην εξωτερική της πολιτική και αυτό ισχύει και για την πολιτική της άμυνας επίσης. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι ε, εξαρτημένη από μη μόνο υπερδύναμη όταν έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αναλάβουμε μόνοι μας την προστασία των δικών μας συμφερόντων. Εδώ και δέκα χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε πάνω από 30 πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς όμως μόνιμες δομές δεν μπορούμε να δράσουμε με ικανοποιητικό τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο ανώτατο στρατηγείο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να, να προσανατολιστούμε και προς κοινούς στρατιωτικούς πόρους που θα γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από την Ένωση με συμπληρωματικό τρόπο φυσικά με το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα αυξήσουμε τη δική μας στρατιωτική παρουσία ότι θα πρέπει να μειώσουμε την διατλαντική μας συνεργασία. Όχι. Σύμφωνα με τα επίπεδα συνεργασίας τα οποία θα προβλεφθούν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να κοστίσει 20 με 100 δις τον χρόνο, ανάλογα με την ευρωπαϊκή συγκυρία. Ε, προφανώς και κάτι θα πρέπει να κάνουμε και σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής άμυνας και η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η αμυντική, θα πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο καινοτόμος. Και γι' αυτό πριν το τέλος του χρόνου θα προτείνουμε την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Η συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στις χώρες που το επιθυμούν να συνδυάσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες στα πλαίσια μιας ενισχυμένης μόνιμης ε, διαρθρωτικής συνεργασίας. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να χρησιμοποιήσουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ κύριε Πρόεδρε αφορά τη λεγόμενη συλλογική μας ευθύνη. Καλό όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό επίσης κάθε χώρα μέλος να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την αντίληψη η οποία λέει ότι η επιτυχία είναι εθνική και η αποτυχία ευρωπαϊκή. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό τότε η κοινή προσπάθειά μας δεν θα επιβιώσει. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει αντικείμενο καλύτερης επεξήγησης. Ζήτησα από τον καθένα από τους επιτρόπους να επισκεφτεί τις επόμενες εβδομάδες τα κοινοβούλια των κρατών μελών και να συζητήσει την κατάσταση της Ένωσης. από την αρχή της εντολής μου οι επίτροποι έχουν επισκεφθεί τα Εθνικά Κοινοβούλια 300 περίπου φορές και θέλω να το κάνουν ακόμα περισσότερο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μόνο αν γίνει πραγματικά κατανοητή. Πρέπει να την εξηγήσουμε καλύτερα. Η Ευρώπη θα γίνει μαζί με τα κρατη και όχι εναντίον των κρατών μελών. Η Επιτροπή της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, θα πρέπει να είναι μια πολιτική επιτροπή, αλλά δεν θα πρέπει ε, να ξεφεύγει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι μια επιτροπή η οποία θα ακούει. Θα ακούει τον πολίτη, θα ακούει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ακούει τα κράτη-μέλη. Και αυτό κάνουμε. Ακούμε το τι θέλουν οι συμπολίτες μας και θέλουμε να το κάνουμε ακόμα και περισσότερο. Μερικές φορές διαβάζω ότι είμαι ένας φυλακισμένος στο μέγαρο του Μπερλεμό και δεν επικοινωνώ με αυτούς τους οποίους υποτίθεται κυβερνώ σε εισαγωγικά. Είμαι ένας γραφειοκράτης καλοπληρωμένος που δεν κοιτάω το τι κάνουν οι άλλοι. Ενώ εγώ σε επίπεδο πολιτικό επικοινωνώ σε καθημερινή βάση με τους πολίτες και θα συνεχίσω να το κάνω. Είναι καθήκον μου, είναι καθήκον μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα, επαναλαμβάνει τις προτάσεις της, ε, κατέθεσε αλλά ταυτόχρονα απέσυρε και πάρα πολλές πρωτοβουλίες τα δύο πρώτα χρόνια και ζήτησε να υπάρξει μια επανεξέταση σε βάθος της ισχύουσας νομοθεσίας, συγκεντρώνοντας την προσοχή μας στους τομείς τους οποίους η Ευρωπαϊκή ε, ε, Κοινότητα μπορεί να προσφέρει, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει, να προσφέρει θέμενη αξία σε έναν χώρο όπου η αλληλεγγύη και η επικουρικότητα συνδυάζονται αρμονικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη, τα τεχνοκρατικά, τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν ε, να καταργήσουν τα χρέη του roaming ε, και είναι μια υπόσχεση την οποία θα τηρήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς κάναμε και μια πρόταση για τα συγκεκριμένα αυτά χρέη του roaming το καλοκαίρι το σχέδιο αυτό είχε καλές προθέσεις, ήταν δίκαιο. Σε επίπεδο επίσης τεχνικό ήταν σωστό, αλλά δεν ανταποκρινόταν στις υποσχέσεις οι οποίες είχαν γίνει. Και τις επόμενες εβδομάδες θα σας κάνουμε μια πολύ καλύτερη πρόταση. Όταν ταξιδεύετε στην Ευρώπη με το κινητό σας τηλέφωνο θα νιώθετε παντού στην Ευρώπη σπίτι σας. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαντούμε για τις πράξεις μας απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε αυτούς που μας εκλέγουν. Γι' αυτό πρότεινα να αλλάξω τον κανόνα που είναι παράλογος κατά τη γνώμη μου, που θέλει οι επίτροποι που ε, παρουσιάζονται στις ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να παρατηθούν από τα αξιώματά τους. Ο Πρωθυπουργό και οι Υπουργοί στα κράτη-μέλη δεν ε, εγκαταλείπουν το αξιωμά του όταν κατεβαίνουν σε εκλογές. Δεν θα πρέπει να το κάνουν και οι επίτροποι. Αν θέλουμε μια επιτροπή υπεύθυνη κοντά στους πολίτες θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ε, επιτρόπους να παίρνουν ραντεβού με τη δημοκρατία και με τις εκλογές, με την καθολική ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, είμαι τόσο νέος όσο το ευρωπαϊκό σχέδιο που το Μάρτιο του χρόνου θα γιορτάσει τα 60 του χρόνια. Ε, είμαι λίγο πιο γέρος εγώ. Έζησα αυτή την ιστορία. Αφιερώθηκα σε αυτήν όλη μου τη ζωή. Από πεποίθηση. Χωρίς δισταγμούς. Ο πατέρας μου πίστευε στην Ευρώπη. Πίστευε στην υπηρετική σταθερότητα, στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην ευρωπαϊκή πρόοδο την κοινωνική ευρωπαϊκή πρόοδο. Ήξερε πόσο πολύτιμη ήταν και πόσο εύθραυστη ήταν η ειρήνη στην Ευρώπη, γιατί πολέ, πολέμησε, Χωρί να το θέλει, χωρίς να το θέλει η χώρα του επίσης. Πιστεύω στην Ευρώπη γιατί ο πατέρας μου μου μεταλαμπάδευσε αυτές τις αξίες και εγώ με τη σειρά μου στα παιδιά μου και εμείς στα παιδιά μας. Τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας σαν κληρονομιά. Μια ένωση η οποία ξεχαρβαλώνεται, που ξέχασε το παρελθόν της, που δεν έχει κανένα όραμα για το μέλλον. Τα παιδιά μας, κυρίες και κύριοι, αξίζουν κάτι καλύτερο. Αξίζουν μια Ευρώπη η οποία θα διατηρεί τον τρόπο ζωής μας και τους που τα υπερασπίζεται, που τα προστατεύει. Είναι και, και η ώρα εμείς οι πολίτες. Τα θεσμικά όργανα, οι κυβερνήσεις, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, να οικοδομήσουν αυτή την Ευρώπη και να την οικοδομήσουμε μαζί. Ναι, ξέρω ότι γίνονται συζητήσεις. Μεγάλες συζητήσεις για την Ευρώπη. Ανάμεσα στους αισιόδοξου φιλοευρωπαίους και στους απεσιόδοξους κατά της Ευρώπης. Αλλά η Ευρώπη έχει τη δική της αποστολή. Τη δική της αποστολή και στον κόσμο. Αλλά ανάμεσα στην απεσιοδοξία που βλέπει μόνο ταμείων και στην αισιοδοξία που τα βλέπει όλα ρόδινα υπάρχει θέληση. Υπάρχει η θέληση η αυτών που δεν κλαίγονται, που δεν εγκαταλείπουν, που δεν παρατάνε τα όπλα και που έχουν στο μυαλό τους και τη μοίρα αυτών που θα μας ακολουθήσουν, τις επόμενες γενιές. Επίσης, ε, μας ενδυναμώνει η θέληση των πατέρων μας. Κάνω έκκληση σε αυτή τη θέληση για να ξεπεράσουμε τις διαιρέσεις μας η ιστορία δεν θα κρατήσει στη μνήμη τα ονόματά μας, αλλά θα κριθεί η δύναμη τη θέλησή μα και των πεπιθήσεών μα. Και τα δύο αυτά θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά. Η ιστορία δεν θα θυμηθεί τον καθένα από εμά, αλλά θα θυμηθεί τα λάθη μα. Α μην κουβαλήσουμε αυτή την ενοχή που θα θέσει τέλο στο ευρωπαϊκό όνειρο. αυτό το βέβαια είναι Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον λόγο θα λάβει τώρα για την ομάδα του ΕΛΚ ο Πρόεδρος κύριος Βέιμπερ. Παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Brexit έκανα λόγο για τη νέα γενναία της ε, Μεγάλης Βρετανίας που θέλει η νέα γενναία αυτή να ανήκει στην Ευρώπη. Σήμερα πάλι θέλω να μιλήσω για τη νέα γενναία ξανά ένα εξαιρετικό καλοκαίρι πέρασε. Πάνω από ένα τέταρτο εκατομμυρίων Ευρωπαίων διαδήλωσαν υπέρ της Ευρώπης. Πήραν τα τρένα του Interrail. Δεν αναζωπήρωσαν την δυσπιστία. Με τους άλλους Ευρωπαίους συνένωσαν τις προσπάθειές τους και από τα μέσα όπως το Σπίγκερ υπήρξαν συνεντεύξεις αυτών των νέων ένας από αυτούς τους νέους, Σέιν είπε ότι ναι, ψηφίσαμε να παραμείνουμε και είναι πραγματικά τρομερό το ότι βρισκόμαστε τώρα εκτός Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ένας νέος Ιταλός, ο Ματέο, ρωτήθηκε ποια ευρωπαϊκή εθνικότητα, εθνότητα δεν θα άντεχε και ποια χώρα δεν θα έπρεπε να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακούστε, η απάντησή του ήταν Καμία φυσικά. Ηλίθια η ερώτηση αυτή. Αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η ατμόσφαιρα μεταξύ της νέας γενναίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν να διαμορφώσουν ένα κοινό μέλλον οι νέοι. Και ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα του Ζαν Κλοντ Juncker σήμερα, στον λόγο που εξεφώνησε. Το μήνυμα για όλους μας. Νομίζω, Ζαν Κλοντ Juncker, με τη σημερινή σου αυτή ε, ομιλία ήταν εξαιρετική η δουλειά σου υπέρ της Ευρώπη και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τώρα, σε σχέση με τους 12 επόμενους μήνες, στρέφομαι σε αυτούς, οι, άνθρωποι στην Ευρώπη δεν θέλουν μια διχασμένη Ευρώπη. Θέλουν να μεριμνήσουμε να υπάρξουν λύσεις, να επικεντρωθούμε σε αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα η Ευρώπη και να μην αναμειγνιόμαστε επί παντός του επίστητου. Και εδώ τίθεται τώρα το θέμα στη συζήτηση, η προάσπιση, η υπεράσπιση της Ευρώπης με ασφάλεια. Γι' αυτό ναι, υπέρ μιας κοινής ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων στην Ευρώπη και μια ασφάλεια των συνόρων που θα μας προστατεύει όλους. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, European Way of Life, έχει αξία για μας. Θέλουμε την ταυτότητα της Ευρώπης, ε, τις ρίζες ε, στον ε, εβραϊσμό και στον χριστιανισμό να τις διαφυλάξουμε. Και θέλουμε μια Ευρώπη ανεκτικότητας. Ευρώπη αλληλεγγύης, οι πλούσιοι να βοηθούν τους φτωχούς. Και στο πλαίσιο της, της κρίσης μετανάστευσης να μην αφήσουμε την Ελλάδα και την Ιταλία μόνες τους, να μην τις εγκαταλείψουμε. Ναι, ένα νέο πρόγραμμα για επενδύσεις. Και ναι, πολλές νέες επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη η European Way of Life, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, είναι για την ευρωπαϊκή κοινωνική αγορά και οικονομία. Και γι' αυτό ευχαριστούμε από την ομάδα μας θερμά, Jean-Claude Juncker και την αρμόδια επίτροπο, ότι τώρα τα θέματα για το διαδίκτυο περνάνε στο προσκήνιο και θα κληθούν τώρα οι εταιρείε ε, να καταβάλουν φόρους. Ευχαριστούμε γι' αυτό. European Way of Life, ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, είναι υπέρ της ανάπτυξης. Μόνο όταν έχουμε καλές προοπτικές για τις εξαγωγές και εξάγουμε τότε μπορούμε μόνο να δώσουμε στους νέους της Νότιας Ευρώπης θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό λέει η δική μου ομάδα ναι υπέρ της ΣΕΤΑ, υπέρ της Συμφωνίας για το εμπόριο με τον Καναδά. Ευρωπαϊκή ταυτότητα και ε, προοπτική για ε, τον επομισμό των ε, δαπανών. Δεν πρέπει λοιπόν τα παιδιά μας να χρωστάνε από τα χρέη τα οποία έχουμε συνάψει εμείς. Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Η Τουρκία είναι σημαντικό εταίρο. Θέλουμε τη φιλία με την Τουρκία. Πιστεύουμε όμω ότι δεν μπορεί να είναι πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα λειτουργήσει αυτό. Και ο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή είναι υπέρ τη δημιουργικότητα. Γι' αυτό ευχαριστούμε για τι προτάσει copyright, για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δημιουργικότητα να προστατεύεται και στην ψηφιακή εποχή. Και ίσω ίσως επιτρέψτε μου στο τέλος αυτή των χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής ε, ζωής, του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, να πω κάτι, μια και ανέφερα το Interrail η καλύτερη ευκαιρία δίνοντας ε, στους νέους ε, των 18 ετών ένα εισιτήριο Interrail από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να βιώσουν την Ευρώπη για τρεις εβδομάδες. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι αυτά τα οποία έχουμε υπόψη να πράξουμε τους επόμενους 12 μήνες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και μια δεύτερη συζήτηση ενώπιον μας στην Πρατισλάβα. Θα έχουμε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εδώ θέλω να απευθύνω μια έκκληση μια έκκληση που θέλω να υπογραμμίσω και αυτή είναι η παράκληση επιτέλους σταματήστε να, ε, να, να ε, δημιουργείτε προβλήματα μεταξύ σας ε, και να έχετε διχογνωμίες πρέπει να είμαστε ενωμένοι αγαπητοί συνάδελφοι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα θέλω να επιλέξω από όλα σε αυτή την νομοθετική περίοδο σε αυτή την νομοθετική περίοδο το Συμβούλιο 148 νομοθετικές ψηφοφορίες ε, διεξήγαγε. 148 νομοθετικές ψηφοφορίες. Η Γαλλία μία φορά πήχε και κατά, κατά τα άλλα πάντα υπερψήφιζε. Η Σεχία και η Πολωνία, η Πολωνία η κυβέρνηση μόνο μία φορά στράφηκε κατά μιας απόφασης του Συμβουλίου και κατά τα άλλα πάντα υπεψήφιζε Οι συνάδελφοι της Ιταλίας πάντα υπερψήφιζαν, ποτέ δεν απήχαν, ποτέ δεν καταψήφισαν. Γι' αυτό η πιο σημαντική παράκλησή μου προς το Συμβούλιο είναι επομιστείτε επιτέλους τις ευθύνες σας, εξηγήστε στους πολίτες σας ε, τι ε, αποφασίζετε στην Ευρώπη, σταματήστε πια με αυτό το φθηνό λαϊκισμό. Ευχαριστώ οι πολιτικοί. πρέπει να έχουν την φλόγα, φλόγα πεποίθησης, φλόγα αρχών και αξιών για αυτά που είναι σημαντικά και πρέπει να πράξουν. Και αυτή ακριβώς αυτός ο ενθουσιασμός που βρίσκεται, βρίσκεται στους νέους. Από αυτούς μπορούμε να μάθουμε. Από τη νέα γενεά της Ευρώπης. Ξέρουν την αξία και αυτής της κοινοτικής κοινή Ευρώπης. Και ας δοθεί μάχη λοιπόν καθημερινά για αυτή την Ευρώπη και έτσι θα το καταφέρουμε από κοινού να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Για τους σοσιαλδημοκράτες θα λάβει τον λόγο ο πρόεδρος κύριος Πιτέλα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, υψηλού επίπεδου η ομιλία του Πρόεδρου Γιούνκερ. Ήταν σοβαρή ομιλία, υπεύθυνη ομιλία. Μας μίλησε και για τα μετά το Brexit, μας μίλησε για το πρόγραμμα των επενδύσεων, το Ταμείο των Επενδύσεων. Είπε πράγματα που ήταν θετικά, δεν μίλησε για τη λιτότητα και τον ευχαριστώ γι' αυτό, μίλησε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πρότεινε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για τους επόμενους 12 μήνες, πράγματι κρίσιμους για τους πολίτες μας. Εμείς θα τον υποστηρίξουμε, θα τον υποστηρίξουμε με θετικό τρόπο, για να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε, να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε. Στην ομιλία σας βρίσκω στοιχεία αντίδρασης στην κατάσταση τη σημερινή. Μετά από τα Brexit άκουσα πάρα πολλά άσχημα πράγματα από τους ηγέτες που έλεγαν είμαστε στην άκρη του κρυμνού, δεν έχουμε ελπίδες πια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία ήταν σαν υπνοβάτες και η Τερέζα Μέη μπροστά σε αυτό το ξεκάθαρο αλλά θλιβερό αποτέλεσμα για μας, ε, συνεχίζει τρεις μήνες μετά να λέει ότι φταίει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τραγικό, είναι γελίο. Εμείς συνεχίσαμε λοιπόν την πολιτική μας ε, και σε οικονομικό επίπεδο ε, υπάρχουν θετικά στοιχεία Δυστυχώς όμως μας προξενούν αλλεργία οι τελευταίοι πρωταθλητές της λιτότητας, ο Υπουργός Σόιμπλε και οι φίλοι του. Νομίζω ότι αυτός ο τυφλός φανατισμός δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εμείς η ομάδα μας είναι μια προοδευτική ομάδα και δεν δέχεται τέτοιου είδους αντιλήψεις. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε μεταξύ μας, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους φιλοευρωπαϊστές σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο, με συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους για να ξεπεράσουμε τους εθνικισμούς και σε εισαγωγικά πατριωτική μορφή της δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι πρώτον αηφόρος ανάπτυξη καταπολέμηση της διαφθοράς, αλληλεγγύη. Ε, νομίζω ότι αυτές οι αξίες είναι συμβατές με τις δικές μας σοσιαλιστικές αξίες. Είμαστε υπέρ των προσπαθειών για το πρόγραμμα επενδύσεων. Θα πρέπει να στηρίξουμε και πιο ρηψοκίνδυνες επενδύσεις. Είμαστε υπέρ της πιστοτικής ένωσης Είμαστε υπέρ της ενίσχυση του Ταμείου για την καταπολέμηση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Ε, είμαστε ε, επίσης υπέρ της σωστής και δίκαιης εφαρμογής ε, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της ύπαρξής της. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε τα μέσα για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Δεν θα πρέπει εμείς να τιμωρήσουμε την Ισπανία και την Πορτογαλία. Δεν θα πρέπει να σταθούμε σαν τον προκρούστη ο οποίος θα τιμωρεί με αυτούς με τους οποίους διαφωνεί. Πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη, πρέπει να στηρίξουμε τον πολίτη που έχει ανάγκη. Αυτά μας τα είχε πει και ο Ζακ Ντελόρ. Θα πρέπει επίσης να καταστήσουμε ηθική την οικονομική δραστηριότητα, καταπολεμώντας τις φοροαποφυγές και φοροδιαφυγές. Θα πρέπει να πληρώνονται οι φόροι εκεί όπου βγαίνουν τα κέρδη. Δεν μπορεί ένας φούρναρης στο Στρασβούργο να πληρώνει περισσότερους φόρους από μια αμερικανική ε, ε, ε, πολυεθνική εταιρεία Θέλουμε επίσης και ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς για τους επιτρόπους και τέος επιτρόπους. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την εγγύηση για τους νέους. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει να σεβαστούμε αυτά που είπατε κύριε Γιούνκερ για το κοινωνικό ντάμπινγκ γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα τέτοιο κοινωνικό ντάμπινγκ και πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Και τέλος Πρέπει να προωθήσουμε την οδηγία για τις προσωρινές μορφές απασχόλησης ε, και για την μετανάστευση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η Φεντερίκα Μογκερίνη είναι μια πραγματική υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε με το σύμφωνο για τη μετανάστευση για την Αφρική. Είναι επαναστατική η πρόταση αυτή και επίσης να βρούμε μια λύση για τους συνόδευτους ανηλίκους, για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, για την ένταξη της Κροατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σέγγεν. Έχετε λοιπόν κύριε Πρόεδρε την δυνατότητα και την ικανότητα να προχωρήσετε στην επόμενη φάση. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο εμπόδιο μπροστά μας, τον φόβο. Δεν πρέπει όμως ο φόβος να μας αποτρέψει από τον στόχο μας. Δεν πρέπει να εμποδίσουμε τους νέους να ζήσουν την Ευρώπη. Πρέπει να παραμερίσουμε τον φόβο με αποφασιστικότητα και να δείξουμε την μεγάλη ευρωπαϊκή μας καρδιά. Ευχαριστώ, Τζάνι. Τον Ιούνιο φέτος ο Βρετανικός λαός ψήφισε να εξέλθει η χώρα του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όσους είναι δυσαρεστημένοι πρέπει να σας πω ότι δυσαρεστημένοι δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν τα σημάδια και σε άλλες χώρες. Και αν συνεχίσουμε να τα αγνοούμε, μην σας εκπλήξει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Το ECR, η ομάδα την οποία ε, ηγούμε, έχει ε, μέλη από 18 κράτη-μέλη που θέλουν ότι είναι καλύτερο για τους ψηφοφόρους και τις χώρες τους. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι έχει βαλτώσει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα πρέπει να γίνει μια επανακίνηση. Αυτά μα λέτε. Αυτά μα τα λέτε κάθε χρόνο. Περισσότερη στρατιωτική ολοκλήρωση. Περισσότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη. Περισσότερο χρέο για τα αυριανά παιδιά. Ούτω ώστε οι σημερινοί σοσιαλιστές να είναι ικανοποιημένοι. Όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Όσο χτίζεται περισσότερη η Ευρώπη, τόσο πιο πολύ θα απομακρύνονται η Ευρώπη. Όσο περισσότερο διαδίδεται τον ευρωπαϊκό υπερεθνικισμό, τόσο περισσότερο θα διωγγώνεται ο εθνικισμό στα κράτη-μέλη. Όσο περισσότερο καταδικάζεται τον ευρωσκεπτισμό, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε ένα πρόεδρο Λεπέν. Και ξέρετε ότι αυτό τους περισσότερους μας φοβίζει. Αλλά αυτές τις ανησυχίες τους, ε, των ανθρώπων τις αγνοείτε και στέλνετε τον κόσμο στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Το θέμα δεν είναι οι ευρωσκεπτικιστέ εναντίον αυτών που θέλουν την ολοκλήρωση. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι να ζούμε σε ασφάλεια, να έχουμε θέση απασχόληση και να έχουμε ευκαιρίε για τους πολίτες μας. Η ομάδα μου, το ECR, πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερη συνεργασία χωρίς περισσότερη συγκεντρωτικότητα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει λιγότερα αλλά καλύτερα. Η επόμενη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να βλουστεύσει αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχει ευελιξία την ευελιξία ενός ε, δικτύου παρά την ε, μονολυθικότητα ενός μπλοκ πολυμορφία και αμοιβαία αναγνώριση αμφισβητείται από το μάντρα της εναρμόνισης που το κοπανάμε ξανά και ξανά. Φορολογική εναρμόνιση, εναρμόνιση, εναρμόνιση. Πολυμορφία σημαίνει επίσης ότι αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρες το ίδιο. Όμως, μερικές φορές σήμερα κάποιες χώρες αντιμετωπίζουμε σαν πιο ίσες από άλλες. Η Γαλλία ξεφεύγει από τους αυστηρούς δημοσιογραμμικού κανόνες γιατί είναι η Γαλλία. Η κυρία Μέρκελ αμφισβητεί κάθε κανόνα για τη μετανάστευση. Οι χώρε στην Ανατολική όμω Ευρώπη ε, και την Κεντρική Ευρώπη στυλιτεύονται από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Και ενώ λοιπόν αγνοούμε του κανόνε, πώ θέλετε να δρούμε με καλή πίστη. Χρειαζόμαστε δημοκρατία. Χρειαζόμαστε ανοιχτό πνεύμα. Και αυτό θα πρέπει να πρετανεύσει και εδώ, σε αυτή την αίθουσα και στα θεσμικά μα όργανα. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η μεγάλη συμμαχία όπου πέντε άντρες από τέσσερις χώρες παίρνουν τις αποφάσεις. Θα ήθελα να τους υπενθυμίσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 751 ε, ευρωβουλευτές και 8 πολιτικές ομάδες και θα πρέπει να τους σεβαστείτε όλους. Η ομάδα μου και οι χώρες που εκπροσωπώ 18 χώρες Θέλουμε η Ευρώπη να πάει σε μια νέα κατεύθυνση, να υπάρξουν σοβαρέ μεταρρυθμίσει. Μεταρρυθμίσει που δεν θα θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλε τι απαντήσει. Μεταρρυθμίσει οι οποίε θα προωθήσουν επιχειρηματικότητα που κάποτε έκανε την Ευρώπη σπουδαία. Μεταρρυθμίσει που θα μα βοηθήσουν να ανταγωνιστούμε, να δώσουμε ευκαιρίε για του πολίτε μα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Για του ε, φιλελεύθερους, ο πρόεδρο τη ε, κύριο Φερχόφστατ, Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Αν κατάλαβα σωστά την τελευταία παρέμβαση, είπε ότι η πηγή του εθνικισμού και του λαϊκισμού είναι λέει εδώ. Εμείς είμαστε λέει η πηγή του λαϊκισμού και του εθνικισμού. Αν κάποιος είναι υπέρ της Ευρώπης, αν είναι κάποιος υπέρ της Ευρώπης, αν κάποιος είναι υπέρ του ευρωπαϊκού οράματος και υπέρ του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ε, τότε κατηγορείται σήμερα ότι είναι η πηγή, λέει, εθνικισμού και προστατευτισμού. Είναι γελίο, παράλογο, αγαπητοί φίλοι, να ακούει κανείς μια τέτοια κατηγορία. Γελίο αφενός, όμως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αφετέρου. Τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, διότι σε ένα θέμα έχει δίκιο ο κύριος Καμάρ η, ανά, η ε, ε, άνοδος ε, του εθνικισμού και του λαϊκισμού είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα πρόβλημα και για την Ευρώπη που θα πρέπει να βρει τις λύσεις. Αληθεύει, είναι, είναι υπέρ της Ευρώπης και από την άλλη πλευρά υπάρχουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που δεν θεωρούν πλέον ότι την Ευρώπη ως την λύση. Και αυτό είναι η πραγματική κρίση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο διχασμός μεταξύ των γενεών θα μπορούσε κανεί να πει. Μεταξύ των νέων που έχουν εμπιστοσύνη και πιστεύουν στην Ευρώπη του μέλλοντος και των άλλων που έχουν τεράστια προβλήματα με αυτή την Ευρώπη. Και γιατί έχουν προβλήματα με την Ευρώπη να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτό. Όχι την νέα ε γενεά, το άλλο τμήμα του πληθυσμού. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό σε μια κατάσταση όπου συζητούμε την κατάσταση τη Ένωση. Έχουν την εντύπωση οι πολίτε ότι δεν ελέγχουν πλέον τη ζωή του ε, και δεν, ελέγχονται, δεν ελέγχεται η ζωή του από του πολιτικού που έχουν εκλέξει ούτε στο εθνικό επίπεδο ούτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό που βλέπουν είναι τρομοκρατία, φοροδιαφυγή, διεθνέ έγκλημα, διεθνή εγκληματικότητα, ροέ μεταναστευτικέ, μεταναστευτικά προβλήματα και δεν προστατεύονται από όλα αυτά από ό,τι βλέπουν το αντίθετο, βλέπουν ανταγωνισμό, ελεύθερες αγορές, ελεύθερο εμπόριο και πηγές αδικίας και ανισότητας αντί ο ανταγωνισμός, το ελεύθερο εμπόριο και τα να είναι μια πηγή νέων ευκαιριών και μια δυνατότητα να εξευρεθεί, να δημιουργηθεί πρόοδο στο μέλλον. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Και μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που υπάρχει αυτό ο διχασμός μεταξύ των γενεών και μεταξύ εκείνων που έχουν χάσει τον έλεγχο τη στη ζωή του, όπω πιστεύουν και δεν θεωρούν ότι εμεί οι πολιτικοί έχουμε την ικανότητα να ελέγξουμε τα πράγματα σε σχέση με τη ζωή του, ε, σε ένα τέτοιο περιβάλλον υπάρχει αν, αναδύεται ο εθνικισμό και ο λαϊκισμός ε, και με τον κύριο Τραμπ στη ΣΥΠΑ. Εδώ έχουμε δικούς μας λαϊκιστές, την κυρία Λεπέν, τον κύριο Μελονσόν. Δεν βλέπω διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστεράς καμιά φορά. Και όλοι έχουν την εξή κατήχηση, το εξής μήνυμα να δημιουργήσουν λέει ένα μεγάλο πλαίσιο ασφάλειας. Λένε ότι με τύχη, με σειρματοπλέγματα μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα και να κρατηθούν τα προβλήματα εκτός Ευρώπης. Ότι δηλαδή οι φράκτες, ε, τα σειρματοπλέγματα μπορούν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Τη μετανάστευση, τις κλιματικές αλλαγές ε, με φράκτες και σειρματοπλέγματα Μα πώς γίνεται να κρατηθούν οι κλιματικές αλλαγές εκτός συνόρων ε, με φράχτες και συρματοπλέγματα όταν βλέπουμε ότι εδώ και σε σχέση με αυτά τα προβλήματα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική. Και τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με υπερεθνικές πολιτικές και υπερεθνικά μέσα και εργαλεία στο μέλλον. Όμως αληθεύει εγώ πιστεύω ότι αληθεύει ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η οργή και ο φόβος των πολιτών δημιουργείται από, αυτή την, από αυτό το διχασμό, από αυτή τη ρήξη. Αφενός έχουμε την παγκοσμιοποίηση που ισοπεδώνει τα πάντα. Από την άλλη πλευρά δημοκρατικές πολιτικές που μόνο σε ένα επίπεδο εθνικό ή τοπικό ε, μπορούν να ε, αναπτυχθούν για να πείσουν και πιστεύω ότι αυτό ήταν και το αίτιο για την ε, χρηματοοικονομική κρίση του 2008 διότι η παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν σταματά και μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα κράτη και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αν θέλουμε να δώσουμε μια θετική απάντηση στις φοβίες, στους φόβους των πολιτών και να κερδίσουμε τον έλεγχο όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις ζωές τους, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις, ευρωπαϊκές προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιορίζουμε με αστυνομευτικά μέτρα τις ε, εθνικές πολιτικές και τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα θα μπορούσε κανείς με μια λέξη να το πει αυτό. Δεν είναι η πηγή αυτών η Ευρώπη, αλλά είναι το αντιστάθμισμα, το αντίβαρο σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση και τα προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και το καρκίνωμα του εθνικισμού και του λαϊκισμού, το οποίο μαστίζει την Ευρώπη. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω εγώ, πρέπει να κάνουμε τη σωστή ανάλυση και νομίζω ανταποκριθήκατε σε, σε αυτό κύριε Γιούγκερ με έναν κατάλογο συγκεκριμένων προτάσεων. Τριών προτάσεων. Πρώτα απ' όλα τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Άμυνας. Επιτέλους ε, θα έλεγα η πρώτη φορά από δεκαετίες που από, την από τη Γαλλική ε, Εθνοσυνέλευση είχε αυτό προταθεί τώρα ε, αναγνωρίστηκε εκείνο το οποίο έγινε το 1954 και υπάρχει μια νέα ε, ε, πορεία και για τις προσπάθειες ε, που έγιναν, για τις προτάσεις που έγιναν σε σχέση με τους Ούγγρους και τους Πολωνούς. Να το κάνουμε αυτό. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν είναι οι Αμερικανοί πια στο μέλλον που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ασφάλειά μας. Εμείς πρέπει να επιληφθούμε των ευθυνών μας γιατί διαφορετικά κανείς δεν θα ενδιαφερθεί για τη γειτονιά μας και την ασφάλειά μας. Και δεν έχω καμία αυταπάτη πρέπει να πω σε σχέση με την απροθυμία αυτών να πορευθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, μια αυθεντική διακυβέρνηση για το ευρώ και την ευρωπαϊκή οικονομία. Είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, Τζάνι Πιτέλα, αυτό που κάναμε μέχρι σήμερα για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που λένε κάποιοι ναι να εφαρμοστεί, κάποιοι άλλοι όχι, να μην το τηρήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Η Γαλλία έχει ένα πρόβλημα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και δεν το τηρεί. Η Γερμανία από την άλλη πλευρά πάλι ε, από τη δική της πλευρά κάποια πράγματα δεν τα τηρεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Σας εθαρρύνω κύριε Γιούγκερ να προχωρήσετε με την έκθεση των πέντε προέδρων, με, του, με την, ε, τον Υπουργό Οικονομικών, με το, ε, τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουμε. Διότι αυτό το παιχνιδάκι με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν μπορεί πια να συνεχιστεί. Θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία, θα γελιοποιηθούμε έναντι εκείνων που παρατηρούν το τι συμβαίνει. Και για την μετανάστευση και την πολιτική ασύλου πρέπει να κινηθούμε όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και την δυνατότητα να το κάνουμε και να υπάρχει η προτροπή ενθάρρυνση να προχωρήσουμε. Το θετικό περιβάλλον είναι δεδομένο. Α κοιτάξουμε και ας δούμε τι έγινε με τον Brexit. Το Brexit ε, δεν είναι ε, πλέον ε, μια, μια επιβάρηση και μια ευκαιρία διαγράφε, αναδύεται εδώ. Γιατί είναι μια ευκαιρία, γιατί θέλει η Βρετανική κυβέρνηση από το Brexit να οδηγηθεί σε μια ευκαιρία και μια επιτυχία. Καθήκον τους είναι και δικό μας καθήκον και δική μας ευθύνη είναι από το Brexit να οδηγηθούμε και εμείς σε μια επιτυχία για την Ευρώπη. Για όλους τους πολίτες της Ευρώπης παρακαλώ. Και είναι μια ε, δυνατότητα αυτή να σταματήσει η δραματική περίπλοκη αποτελμάτωση των ε, θεσμικών μας οργάνων. Και θέλω να ολοκληρώσω. Το Brexit δεν είναι θέμα ποινών και κυρώσεων. Δεν είναι θέμα αντεκδίκησης και εκδίκησης. Είναι, όπως το βλέπω εγώ, το Brexit ένα θέμα μιας σωστής, σωστού συσχετισμού μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρώπης και πέρα και πάνω από αυτό είναι για το πώς επιθυμούμε εμείς την Ευρώπη να τη διαμορφώσουμε, τη δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αυτό είναι το πρόταγμα, το διακύβευμα και αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση για το, ε, την κατάσταση της Ένωσης και το μέλλον. Ας σταματήσουμε σε αυτό το σημείο στις δύο όχθες ε, ένθεν και ένθεν ε, της μάχης μεταξύ Βρετανίας και Ευρώπης. Πρέπει να επανεπινοήσουμε την Ευρώπη και να προχωρήσουμε προς αυτήν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, το είδα, το είδα. Ε, κύριε Φερχόφστατ, ο κύριος ε, Μπέτεν ανήκει στην ομάδα που όλο αυτό το ε, χρόνο παραπονείται για τις υπερβάσεις χρόνου των αγορητών. Τώρα θέλει να θέσει μια ερώτηση. Συμφωνείτε. Παρακαλώ κύριε Μπέτεν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριε Φερχόφστατ, καταρχάς συγχαρητήρια για το νέο διορισμό σας σαν διαπραγματευτή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Brexit. Εγώ πάντα με χαρά σας ακούω, είστε λογικός, συνεκτικός αυτά τα πιστεύω σας. Θεωρείτε ότι η Ευρώπη πρέπει να ορμήσει προς τα εμπρός έτσι κι αλλιώς ε, θα υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ μας, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, ξέρουμε τα ε, πιστεύω σας. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα πρέπει να επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο το ταχύτερο δυνατόν. Το 50 είναι κάτι το μακρόχρονο, κάτι το μη απαραίτητο. Μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ έγραψα και ένα βιβλίο για το πώς ε, θα πρέπει να γίνει ε, ο διαχωρισμός το ταχύτερο δυνατόν. Θα σας το δώσω μετά τη συνεδρίαση. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπότεν για την θετική αξιολόγησή του του διορισμού μου. Είναι πρώτη φορά που το ακούω αυτό από τη δική του πλευρά. Και να του πω επίσης ότι ναι, θέλω γρήγορα. Συζητήσατε τον λόγο για διαδικαστικό. Ισούλη, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με την τήρηση του χρόνου, λέει ο Σούλικ. Σε άλλες περιπτώσεις ε, χτυπούσατε με το κουδουνάκι το σφυράκι. Θα το κατανοούσα αυτό, θα το χαιρέτιζα αν είχαμε τον, τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλους τους αγορητές. Κύριε Σούλικ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Σούλικ, δεν ξέρω πόσο συχνά είσαστε στην Ολομέλεια όταν εγώ προεδρεύω τη Ολομέλεια. Τι περισσότερε φορέ ασκούνται επικρίσει ότι δεν τηρώ τα χρονικά όρια των αγοριτών. Και σε εσά ε, κιόλα. Επειδή είμαι πεισμένο ότι σε μια τέτοια συζήτηση αρχηγοί πολιτικών ομάδων ε, που για παράδειγμα σε σχέση με του εργατικού ή τον κύριο Πιτέλα που ομιλούν εξ ονόματο ε, εκατοντάδων βουλευτών χρειάζονται σίγουρα κάποια λεπτά παραπάνω σε μια τέτοια σημαντική συζήτηση. Αυτό ισχύει για όλου του αρχηγού ομάδων και πολιτικών ομάδων, κοινοβουλευτικών ομάδων. Και είμαι εξίσου δίκαιο και σχέση με την κυρία Τσίμερ για παράδειγμα. Και τώρα στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο η κυρία Τσίμερ ακριβώς. Παρακαλώ. Η κυρία Τσίμερ σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ για το ότι προαναγγέλλετε ότι θα κλείσετε ένα μάτι και θα σας τελέγει γενναιόδωρος πάλι μαζί μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε κάτι εδώ. Περί τίνος πρόκειται. Θέλουμε το status quo να τηρήσουμε με όλα τα ολισθήματα και όλα τα κακό κείμενα αυτά να διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη και στο τέλος να αποτύχουμε ή θέλουμε μια νέα δημοκρατική κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποτολμήσουμε ως το, απο, τόλμημα και ως εγχείρημα, ως διακύβευμα. Εδώ πιστεύω ότι βάθρων πρέπει να εξηγιανθεί το ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα και να μην κάνουμε μερεμέτια. Το ευρωπαϊκό αυτό, ο ευρωπαϊκός οίκος πρέπει να γίνει πάλι κατοικήσιμος και για τους πολίτες πάλι στέγαση με ασφαλή ε, διαμερίσματα με ε, δυνατότητα προοπτικής για το μέλλον για τους νέους, για τη νέα γενεά για την απασχόλησή τους για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης φτώχειας ε, και της, των προβλημάτων κάνουμε όμως πολλά, πολύ λίγα πράγματα και δεν πιστεύουμε σε όλα αυτά πια δεν τα πιστεύουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροτεχνήματα υποσχέσεις που δίνονται λαϊκίστικα. Κανένας δεν είπε ξεκάθαρα ότι η μέχρι τούδε προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στοιχηματίζει δηλαδή στη συνολική ανταγωνιστικότητά της και αυτό να αποβαίνει πάντα εις βάρος των πολιτών στο τέλος τέλος που θα πληρώνουν τα σπασμένα και όλα τα βάρη των χρεών και την επιβάρηση των εθνικών προϋπολογισμών και τις περικοπές των κονδυλίων στον εθνικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες τους ιδιωτικοποίηση δημόσιων κρατικών υπηρεσιών κτλ. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο. Όμως αν δεν αλλάξουμε όλα αυτά, αν δεν αλλάξουμε αυτές τις προοπτικές μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα γυρίζουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Η γάτα θα δαγκώνει συνέχεια την ουρά της. Δεν θα υπάρχει διέξοδος. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Θα υπάρχουν διαρκώ ε, ε, ένα διαρκή εγκυβωτισμό, μια ε, α το πω έτσι πορεία χωρί προοπτική. Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, γιατί έχουμε ανα, αναδυόμενο εθνικισμό και όλο και μεγαλύτερες τάσεις εθνικισμού στα κράτη-μέλη, ε τότε εδώ υπάρχει ένα αίτιο επειδή οι κυβερνήσεις αφεαυτών τους συνεισφέρουν να απλώσουν το κόκκινο χαλί τον τάπιτα αυτό υπέρ τέτοιων εξελίξεων και στο τέλος τέλος να ελαχιστοποιείται η Ευρώπη δίνεται στους ακροδεξιούς, στους ακροδεξιούς λαϊκιστές ε, αυτή η, ας το πω έτσι, δραστηριότητα και πρωτοβουλία. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε και δεν άκουσα το τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτός. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να εκδημοκρατιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει ένα πλαίσιο δημοκρατικής διαμόρφωσής της και εδώ τα πράγματα δυστυχώς δεν υπάρχουν και βλέπουμε σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε, είναι πολλά περισσότερα αυτά που χρειαζόμαστε. Για δείτε για παράδειγμα τις ευθύνη σας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για τους πολίτες. Δεν είπατε, δεν έγινε τίποτα, δεν αναφέρθηκε γι' αυτό. Εδώ λοιπόν για το, ε, τα θεμέλια τα δημοκρατικά δεν κάναμε τίποτα για το πώς θα διαμορφώνεται αυτό το πλαίσιο με τους πολίτες και υπέρ των πολιτών. Δια, διατυπώνω την ερώτηση προς εμάς και εσείς να τη διατυπώσετε στο Συμβούλιο. Βλέπουμε ότι ο προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, για τα ερωτήματα ποιος κυβερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, δόθηκαν τέτοιες απαντήσεις όπως οι λομπιίστες. Δεν είναι λέει δημοκρατικά εκλεγμένοι, τα αιρετά μέλη που εκλέγονται από τους πολίτες για να τους εκπροσωπήσουν. Και δεν επαρκούν όλα αυτά να αναφέρονται σε σχέση με τον Παρόζο και τους λομπίστες. Κάντε κάτι παραπάνω σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής κύριε Γιούγκερ. Κατανοήστε επιτέλους ότι οι πολίτες θέλουν να συμμετάσχουν, θέλουν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να λαμβάνουν τετελεσμένες αποφάσεις ε, ως ε, ε, πραγματικότητα και ως τετελεσμένα γεγονότα άκουσα πολλές φορές να αναφέρεστε σε αυτά τα θέματα. Σε ποιον απευθύνεστε, σε ποιον ζητάτε να ανταποκριθεί. Εσείς πρέπει κάτι να κάνετε ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Συμβούλιο να δράσει για να υπάρξει κάποια βελτίωση. Εδώ είδαμε ότι το Brexit αποφασίστηκε με ένα δημοψήφισμα και τώρα μπορούν να γίνουν λέει, πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν μπορούσαν να, έχουν, να είχαν γίνει. Ε τότε τι κάνουμε. Συζητούμε για μια κοινή ασφάλιση ανέργων. Συζητούμε για κοινού ε, ελάχιστου Ευρωπαϊκού μισθού ε, για του εργαζόμενου. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να διατυπώσετε. Αναμένουμε συγκεκριμένε ερωτήσει και απαντήσει ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά. Κυρία Σίμε, παρακαλώ ολοκληρώστε λέει ο πρόεδρο η κυρία Τσίμερ, παρακαλώ σταματήστε τους αριστερούς να τους εντάσσετε και να τους ευθυγραμμίζετε σε μία γραμμή ε, και να τους ταυτοποιείτε με τους ακροδεξιούς που θέλουν να γύρουν φράχτες και σειρματοπλέγματα. Ευχαριστώ. Για τους πρασίνους θα λάβει τον λόγο η κυρία Πρόεδρος τους, η κυρία η κυρία Ρεμπέκα Χάμς, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα, οτιδήποτε και αν συζητείτε αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κεκτημένα και τα επιτεύγματά της και με τα τροτά της σημεία είναι που τα γνωρίζουμε καλύτερα η καλύτερη απάντηση για τον εθνικισμό μια και εμείς μάθαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 60 χρόνια, σε 6 δεκαετίες, ότι τα συμφέροντά μας από κοινού μπορούμε καλύτερα να τα υπερασπιστούμε και τις αξίες και αρχές μας μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα από κοινού ενωμένοι. Για αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για μας η απάντηση στην ομολογουμένως απειλή της παγκοσμιοποίησης και τους φόβους παγκοσμιοποίησης και για την κυρία Μογκερίνη και για άλλους ε, γιατί ζητείτε μεγαλύτερη αρμοδιότητα στις Βρυξέλλες αλλά όλα έχουν το σωστό χρόνο στον οποίο πρέπει και μπορούν να γίνουν. Είμαι πεισμένη ότι δεν μπορούμε θεσμικές αλλαγές να συζητήσουμε πρώτα και κύρια αλλά σήμερα Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της και να κερδίσουμε αυτή, την, να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Να ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία, την φιλελεύθερη ανοιχτή Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Διότι αυτό είναι εδώ το οποίο πιέζεται και διακυβεύεται μετά από πολλές εξελίξεις ε, των, των τελευταίων τελευταίων ε, αυτών μηνών και ετών. Τι θέλουμε να κάνουμε εμεί οι πράσινοι. Θέλουμε να κινηθούμε προς μια κοινή ευρωπαϊκή πορεία. Πέρυσι ένα μικρό τμήμα των πολιτών που παγκόσμια βρέθηκαν υποδιωγμό και κατέληξαν ως πρόσφυγες και μετανάστες σε εμά Είδαμε τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση με μια τέτοια φυγή παγκοσμίων διαστάσεων, ένα τέτοιο διωγμό και φυγή παγκοσμίων διαστάσεων. Και βλέπουμε ότι όταν έχουμε πολιτικές τάσεις σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσεις και πόλωση που προκαλείται, θέλω να πω εγώ ότι με την ομάδα μου είμαι πεισμένη ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αρθούν στο ύψος των υποχρεώσεων τους και να δεχθούν πρόσφυγες και μετανάστες και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτών των ροών μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών καλύτερα θα προσευχόμουν να μπορέσει να τηρηθεί και να διατηρηθεί η εκεχηρία στην Συρία. Όμως ε, πρέπει να δούμε ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσουμε και να πράξουμε πολύ αποτελεσματικότερα πολλά πράγματα. Και δεν πρέπει εδώ να οδηγούμαστε σε ε, υπεκφυγές. Πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη πολιτική για, τα, για τις χώρες της Αφρικής. Αν δεν έχουμε μια λειτουργούσα, λειτουργική πολιτική για το άσυλο, τα προβλήματα που γνωρίσαμε πρόσφατα θα επανέλθουν και με μεγαλύτερη ένταση και πολύ σκληρότερα. Η αλληλεγγύη. Για την αλληλεγγύη κυρίες και κύριοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακούσαμε πολλά. Απαντήσεις ε, με αλληλέγγυο τρόπο σε σχέση με τη δυστυχία των άλλων όλα αυτά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται ε, ε, ε, με εσωστρέφεια και δεν εκφράζει αλληλεγγύη και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ πόλεων και υπαίθρου όταν έχουμε τεράστια προβλήματα σε σχέση με τις κλινικές, τα νοσοκομεία και τα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν λειτουργεί ε, τίποτα και υπάρχει και τρομοκρατία και υπάρχουν τόσες πολλές πηγές και αίτια για την ε, ε, δημιουργία κλίματος ανασφάλειας. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας εμείς. Με τις απαντήσεις μας δεν μπορούμε να έχουμε τις αυταπάτες ότι χωρίς την προσπάθεια και την συνεργασία των κυβερνήσεων μπορούν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Διότι το πρόγραμμα επενδύσεων που αναφέρατε κύριε Γιούγκερ είναι ναι μεν καλό αλλά ανεπαρκές για να ενδιαφερθεί κανείς για την ανεργία των νέων και να δίνει απαντήσεις στην ανεργία, ανεργία των νέων με εισιτήρια Interrail κύριε Βέμπερ όπως το κάνατε αυτό είναι αναξιόπιστο, είναι γελίο πρέπει κάτι σοβαρότερο να γίνει και για να δούμε το του θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και ε, ε, ανάπτυξης. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ανεργίας των νέων και για τα προβλήματα της, ε, των κλιματολογικών αλλαγών. Αν δεν επικυρωθεί η Συμφωνία των Παρισίων, αν δεν είμαστε αποτελεσματικοί και δεν επενδύσουμε στις ανανεώσιμες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να απελευθερωθεί ένα ολόκληρο δυναμικό που θα φέρει αποτελέσματα υπέρ όλων όλων κυρίες και κύριοι, ως πράσινοι, πάντα είμαστε πρόθυμοι τα κεκτημένα και τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία καταναλωτών, στην προστασία ε, των ψηφιακών δεδομένων, στην ε, προστασία για τα θέματα κλιματολογικών αλλαγών και των κοινωνικών θεμάτων. Αν όλα αυτά τα κεκτημένα και επιτεύγματα θέλουμε να τα υπερασπιστούμε υπέρ των πολιστών και πρέπει να είμαστε σε θέση να το κάνουμε και έναντι της TTIP, διότι αν δεν το κάνουμε θα χάσουμε ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών μας σε τεράστιο βαθμό. Ευχαριστώ. E θα λάβει τον λόγο τώρα για την e ο Ευχαριστώ. Η παράδοση αυτή για αυτή την ετήσια ομιλία ξεκίνησε από τον προκάτοχό σας, τον κύριο Μπαρόζο. Και τώρα είναι καλή ευκαιρία και νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Μπαρόζο για αυτή τη νέα καλοπληρωμένη του δουλειά στην Goldman Sachs. Ε. Όλοι μαζί. Συγχαρητήρια. Αυτό θα συμβεί και με εσά, κύριε Γιούνκερ. Θα σα φροντίσουν ε, οι φίλοι σα τα υψηλά αξιώματα. Ε, με όλα αυτά που άκουσα σήμερα, χαίρομαι που ψηφίσαμε να φύγουμε. Είναι σίγουρα ότι δεν θα μάθετε τίποτα από τον Brexit. Τα ίδια και τα ίδια. Η ίδια συνταγή, περισσότερη Ευρώπη μας κοπανάτε. Και μάλιστα πιο στρατιωτική Ευρώπη. Ευρωπαϊκό στρατό, κοινή άμυνα. Και πολλοί από εσά λέτε ότι η Αμέρικα δεν θα είναι εδώ πια θα πρέπει εμείς να τα καταφέρουμε τις δικές μας στρατιωτικές δομές. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα οικοδόμημα αυτό για την ειρήνη α, η Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι πάτε προς επικίνδυνες οδούς. Δεν πρόκειται να, να, να σταματήσετε τις ε, κεντρικές και ανατολικέ χώρες να πούνε όχι στις ποσοστώσεις της κυρίας Μέρκελ για τη μετανάστευση. Και θα έχετε περισσότερα δημοψηφίσματα να αντιμετωπίσετε. Σε ό,τι αφορά τον Brexit όμως, ίσως έχετε δίκιο που είσαστε λιγάκι επικριτικοί για την Βρετανική κυβέρνηση, που συμφωνώ πρέπει να επιταχύνει λιγάκι να σκουμποθεί. Εσείς όμως συνεχίζετε και έχετε ετοιμάσει τους ε, δικηγόρους για το διαζύγιο. Έχουμε τον Γκί Φερχόφσταντ. Να ο άνθρωπος ο οποίος θα διαπραγματευτεί το Brexit. Εμείς πιστεύαμε ότι ο αυτός ο οίκος είναι ένας ναός, ενώ και ο Φερχόφσταντ είναι ο προθιερέας, ένας φανατικός. Υπάρχει ένας πραγματικός ε, θήκης στην αίθουσα. Αν υπάρχει, είστε εσείς. Γιατί θέλετε σημαίες, ύμνους. Είσαστε ένας Ευρωπαίος εθνικιστής. Και νομίζω ότι αυτή, αυτός ο διορισμός σημαίνει κήρυξη πολέμου σε οποιαδήποτε λογική διαπραγματευτική διαδικασία. Εάν συνεχίσετε με αυτό το δογματισμό ε, που λέτε ότι για να έχουμε ε, μηδενικές ποσοστώσεις εμείς θα πρέπει να δεχτούμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί θα είναι πολύ καλύτερα αυτά που θα έχουμε από τη σημερινή συμφωνία που έχουμε. Για εκατοντάδε χιλιάδες ε, ε, εργαζόμενου Γερμανού στην αυτοκινητοβιομηχανία, όλα αυτά είναι κακά νέα. Γιατί είμαστε μεγαλύτερη αγορά και με την οποία κάνουν εμπόριο πολύ επικερδές παγκόσμια. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι μια κοινή λογική προσέγγιση. Και θα έπρεπε αυτό το κοινοβούλιο να αναγνωρίσει το λάθος του και να βρει κάποιον ο οποίος είναι φίλος του Ηνωμένου Βασιλείου, που του αρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο, για να είναι ο επικεφαλής αυτών των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Äh, Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λεπέν, Μαρίν Λεπέν. Καλημέρα κύριε Γιούνκερ. Ε, καιρό είχα να ακούσω τόσο άνοστη ομιλία. Όραμα πουθενά. Ε, μιλάμε για επίπεδο εγκεφαλογράφημα δηλαδή, τίποτα, μηδέν. Εκτός, εκτός πρέπει να πω βέβαια, εκτός από μια στιγμή εξαιρετικού χιούμορ που είπατε εσείς ότι καταπολεμάτε τις φορολογικές ε, συμφωνίες για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν πήρατε είδηση. Δεν βλέπετε τι θέλουν οι λαοί της Ευρώπης. Θέλουν να ξαναβρούν την ελευθερία τους. Θέλουν να ξαναβρούν την ανεξαρτησία τους στην ουσία εσείς ε, διαβάζετε και ο κύριος Βέμπερ ε, τι λένε οι εφημερίδες. Και έτσι διαβάζοντας αυτά που λένε εφημερίδες πιστεύουν ότι κατάλαβαν το ότι θέλουν λαοί. Όχι, τα αποτελέσματα των εκλογών να βλέπετε. Στους νέους το κόμμα μου στη Γαλλία είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό να βλέπετε. Το Brexit έσπασε ένα ταμπού. Οι Βρετανοί έδειξαν ότι είναι δυνατόν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς όφελός τους. Οι καταστροφικές προβλέψεις εις βάρος τους ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Μια χαρά πάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σοκ το οποίο εσείς θέλατε να δούνε, να δείτε μάλλον την αποκάλυψη η οποία θα χτυπούσε τους Βρετανούς, ξεχάστε τα αυτά. Οι λύσεις τις οποίες προτείνεται δεν αλλάζουν ποτέ. Όλο και περισσότερη Ευρώπη. Και στη γεωργία και στη μετανάστευση και στην οικονομία θέλετε η Ευρώπη να προχωρήσει και να μας προστατεύσει όλους. Κανέναν δεν προστατεύει η Ευρώπη. Είναι λόγια κενά αυτά τα οποία λέτε. Καταργώντας τα εθνικά σύνορα ε, για χάρη του Σέγγεν στην ουσία εποφελείται το οργανωμένο έγκλημα. Επιτίθεστε στην έννοια του κράτους και γι' αυτό ακριβώς οδηγείται στον απομονωτισμό, στον Ισλαμισμό, στην τρομοκρατία. Από τι μας προστατεύει η Ευρώπη, από την ασφάλεια μας προστατεύει η Ευρώπη. Στην ουσία σώζεται το ευρώ καταστρέφοντας τις χώρες του Νότου Διαλύεται τις επιχειρήσεις, έχετε φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο ε, την ανεργία. Από τι μας προστατεύει λοιπόν η Ευρώπη, από την ευημερία μας προστατεύει η Ευρώπη. Οδηγείται σε όξυνση των εντάσεων. Εσείς δείχνετε ότι περιφρονείτε τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Από τι μας προστατεύει λοιπόν η Ευρώπη. Από την ελευθερία μας προστατεύει, από τη δημοκρατία μας προστατεύει. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Η Ευρώπη έχει ανάγκη άλλη από αυτήν που προτείνεται. Μόνο οι εθνικές κοινότητες θα δώσουν τις λύσεις. Αφήστε τα έθνη να απελευθερωθούν. Αφήστε τα να συνεργαστούν μεταξύ τους όπως το θέλουν. Χωρίς Βρυξέλλες. Καλύτερα από τις Βρυξέλλες. Να φανείτε δημοκράτες. Αφήστε τους λαούς της Ευρώπης να είναι κυρίαρχοι της μοίρα τους. Κυρία Ευρωβουλευτά Λεπέν, ο κύριος Κόμπερν, Ευρωβουλευτής, θα ήθελε να διατυπώσει ερώτηση. Τη δέχεστε, συμφωνείτε. Uh, Κυρία Λεπέν, θα ζητήσετε να υπάρξει ένα Brexit να βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εκστρατεία για την Προεδρία που θα κάνετε να πω ότι ακριβώς επειδή σέβομαι την δημοκρατία, το δημοψήφισμα είναι η καλύτερη της έκφραση. Εδώ και τέσσερα χρόνια λέω ότι θα οργανώσω ένα δημοψήφισμα για να μπορέσουν και οι Γάλλοι να αποφασίσουν για την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λάβει τον λόγο τώρα η, μία εγγεγραμμένη κυρία Ντότς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά τη δημοκρατική απόφαση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στις 23 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καθορίσουν και να οικοδομήσουν μια αμοιβαία εποφελή σχέση που θα βασίζεται στη συνεργασία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια και την ευημερία αυτό δεν έχει νόημα μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την ΕΕ. Είμαστε η πέμπτη παγκόσμια μεγαλύτερη οικονομία και η μεγαλύτερη αγορά όσον αφορά τα γερμανικά οχήματα και μεγαλύτερο εισαγωγέα γαλλικών γεωργικών προϊόντων. Μα χρειάζεται λοιπόν η Ευρώπη. Τώρα πρέπει να συνεργαστούμε με ένα νέο τρόπο προ όφελο όλων μα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια μεγάλη χώρα. Θα μπορέσει να ευημερήσει. Η Ευρώπη όμω είναι ο σύμμαχός της. Ε, ας μην αφήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις να τερματιστούν με μια άγωνη αντιπαρά, αντιπαράθεση Υπάρχουν ευκαιρίες λοιπόν και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία υποστηρίχθηκε εδώ σε εγχείρημα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τα χερσαία σύνορά μας θα γίνουν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η πρόοδος η οποία επετεύχθη να απεμποληθεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να στρεφόμαστε και προς την Ευρώπη και παγκόσμια ώστε να μπορέσει να συνεχίσει η ευημερία εκεί όπου η ειρήνη, η δημοκρατία θριάμβευσαν. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε Ντότς, ο κύριος Τένοκ, Ευρωβουλευτής, θέλει να διατυπώσει ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Uh, Northern Ireland, Βόρεια Ιρλανδία πολύ σωστά ψήφισε να παραμείνει, αλλά δυστυχώς η υπόλοιπη χώρα ψήφισε το αντίθετο. Είπατε ότι θα υπάρχει μια ευκαιρία με τα σύνορα ανάμεσα στην Βόρεια Ιρλανδία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Τι θα γίνει με το ε, εμπόριο όμως, ε, με αυτό το σκληρό σύνορο ε, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει προβλήματα σε αυτό το εμπόριο ή όχι. Ireland... Σε ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, ψηφίσαμε να παραμείνει. Αλλά είμαι περήφανη που είμαι τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου και συνολικά το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σέβομαι και θαυμάζω την απόφαση του, των υπόλοιπων συμπολιτών μου. Στη Βόρεια Ιρλανδία έχουμε την εξή κατάσταση. Θα είναι το μόνο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου η Βόρεια Ιρλανδία που δεν έχει ε, χερσαία σύνορα με άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Με, δηλαδή κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα δημιουργήσει ε, προκλήσεις. Ε, θα δημιουργήσει προκλήσεις και για τους ταξιδιώτες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε όμως τα προβλήματα που θα μπορέουν από αυτό το σύνορο. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντότζ. Τώρα, <clears throat> εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος Υπουργός Κόρτσοκ θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Συνήθως ομιλώ από αυτή τη θέση για να εκπροσωπήσω το Συμβούλιο. Θα κατανοήσετε ότι δεν θα είμαι σε θέση να το πράξω αυτή τη στιγμή διότι όλο το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί με βάση τα όσα εξέθεσε ο πρόεδρος Γιούνκερ σε σχέση με τα προγράμματα της Επιτροπής ε, για του χρόνου βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Ε, τον ευχαριστούμε όμως ε, που δημιούργησε μια θετική ημερήσια διάταξη με ένα θετικό θεματολόγιο σε σχέση με την, ε, τον Υπουργό και την ε, ε, παρουσία του όταν παρουσιάστηκε ο λόγος, εκφωνήθηκε ο λόγος για την κατάσταση της έννοιας της Ένωσης. Θέλω να σας διασφαλίσω ότι με επιτακτικό χαρακτήρα κατεπηγόντως πρέπει να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν χρειάζεται εδώ να υπησέθω σε λεπτομέρειες ότι είναι χωρίς προηγούμενο αυτές οι προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να τύχουν ε, γιατί διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το πρώτο θύμα του λαϊκισμού και ο λαϊκισμός δεν επιλύει ε, προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα μόνο. Θα ήθελα να πω τα εξή έχοντας ε, προσέξει τον λόγο του κυρίου Γιούγκερ. Επιβεβαιώνει η Σλοβακική Προεδρία τις αρχές επί των οποίων θεσπίσαμε τις προτεραιότητές μας Θέλουμε να δημιουργήσουμε, να φέρουμε χειροπιαστά αποτελέσματα προ όφελο των πολιτών μα και να σταματήσει ο διχασμό και ο κατακαιρματισμό. Δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι πολλοί αναφέρθηκαν στην επικείμενη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Πρατισλάβα την Παρασκευή. Ποια είναι η αρχική ιδέα που βρίσκεται πίσω από αυτή τη σύνοδο. Είναι πολύ απλή η απάντηση. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνήθαν τον ε, Ιούνιο μετά την ε, αρνητική ψήφο στο δημοψήφισμα για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και πρέπει εδώ σε σχέση με την κατάσταση της Ένωσης να αναζητηθούν οι σωστές απαντήσεις έπρεπε να, ε, τότε να γίνει αυτό η αναζήτηση σωστών απαντήσεων μπορεί να υπάρχουν ε, αποκλίνουσες απόψεις αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην ε, συζήτηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Πρατισλάβα. Θα πρέπει να υπάρχει ο κοινό στόχος να εξευρεθεί κοινό πεδίο για την την εξέβρεση μελλοντικών απαντήσεων στις προκλήσεις και αυτό θα είναι το εγχείρημα στην ε, Μπρατισλάβα. Θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτή την αναζήτηση απαντήσεων και θα έχουμε και την 60η επέτειο ε, ε, του εορτασμού των συνθήκων της Ρώμης και θα πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία της Μπρατισλάβας να προχωρήσουμε. μόνο ένα πρόκληση μετανάστευση. Σας ευχαριστούμε για το ότι αποστεί στείλατε μια έκκληση προς την ε, Σλοβακική Προεδρία για την αναζήτηση λύσεων που θα δώσουν δυνατότητα να υπερβούμε τις ε, επιφυλάξεις κρατών μελών για τα θέματα μετανάστευσης και να δημιουργηθεί μια κοινή βάση για αυτά τα θέματα με βάση την αλληλεγγύη. Ε, δεύτερον, σε σχέση με την ασφάλεια, εσωτερική και εξωτερική, φυσικά θα έχει τεράστια εμβέλεια, τεράστια σπουδαιότητα αυτό το θέμα. Και τέλος, θέλουμε καλύτερα να επικοινωνούμε όσο να και να παρουσιάζουμε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τέλος, η Σλοβακική Προεδρία, Πρόεδρε, για να επιτευχθούν χειροπιαστά αποτελέσματα και να μπορέσουμε να πετύχουμε όσο περισσότερα μπορούμε, η βάση θα πρέπει να είναι η διοργανική συμφωνία. Αυτό θα είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα, θα τονίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την... το σημείωμα την επιστολή προς την Προεδρία και ελπίζω ότι θα μπορέσουν οι Υπουργοί να καταλήξουν σε μια κοινή δήλωση, κοινή διακήρυξη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νομοθετικές προτεραιότητες. Κύριε Πρόεδρε, ήταν προνόμιο για μένα το ότι μπόρεσα να παραστώ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρος. Για το ΕΛΚΑ ο κύριος Ευρωβουλευτής Ρόιλ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστώ πολύ Πρώτον για το ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, μας ε, οδήγησε σε ένα προβληματισμό για τις ε, θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ότι η απάντηση μπορεί να είναι χειροπιαστά αυτά τα οποία μπορούμε να ε, δώσουμε με κάθε προσπάθεια από πλευρά μας. Θέλω να εξειδικεύσω κάτι. Κατά του λαϊκισμού βοηθά όταν έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αξιοπιστία μεγαλύτερη κερδίζουμε όταν δείχνουμε, όταν τηρούμε

κανόνες και αρχές και αξίες. Και γι' αυτό σε σχέση με τα όσα συμφωνήθηκαν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και να τα τηρούμε. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες του παιχνιδιού και θεματοφύλακας όλων αυτών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, να θα κατά των λαϊκισμών. Να έχουμε δικές μας ξεχωριστέ θέσεις για να κερδίζουμε αξιοπιστία. TTIP, Συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ε, ΗΠΑ. Εδώ πρέπει να δούμε ότι διαφοροποιούνται τα πράγματα. Δεν είναι δική μας δουλειά να μπορέσουν τα πράγματα. Ε, πρέπει να πετύχουμε τα πράγματα τα οποία είναι σωστά και αναγκαία να προχωρήσουν. Και οι λύσει ε, δεν είναι μόνο στο επίπεδο διακηρύξεων. Πρέπει να είναι χειροπιαστέ και λειτουργικέ. Αυτό οφείλουμε στου πολίτε μα που αντιμετωπίζουν προβλήματα για την ασφάλεια. Τι κάνουμε λοιπόν για την ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά του πολίτε μα και τη δημιουργία δημιουργία Τι κάνουμε σε σχέση με τα ταξίδια που κάνουν και ξεκινούν και για την ε, επιτήρηση και προστασία των εξωτερικών συνόρων. Δεν χρειάζονται δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτα καινούριο. Αυτά τα οποία έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε περιγράψει πρέπει να τηρούνται. Και τέλος, ε, όποιο θέλει να δημιουργηθεί ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν επαρκεί να υπάρχουν μόνο χρήματα. Πρέπει να δημιουργηθούν όροι και προϋποθέσεις επιχειρήσει να μπορέσουν να δράσουν αποτελεσματικά αποτελεσματικά με έδρα την Ευρώπη. Εδώ τεράστια βήματα πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά πρέπει χρειαζόμαστε ακόμα για να επιτευχθεί αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκε στη συνέχεια παρακαλώ. Yes, Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους πολίτες να ελέγχουν τη ζωή τους, να ελέγχουν τη μοίρα τους. Αυτό σημαίνει καλύτερες λύσεις, αυτό σημαίνει καλύτερες ευρωπαϊκές λύσεις. Εσείς με την ομιλία σας κάνατε θετικές προτάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως θα ήθελε να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας στους τομείς στους οποίους αναφερθήκατε με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο. Ζητάτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πάρει τις απαιτούμενες αποφάσεις στην Πρατισλάβα. Νομίζω ότι στα πλαίσια του οδικού αυτού χάρτη θα πρέπει να τονίσουμε τον κοινωνικό πυλώνα, έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να υπολογίζουν σε κοινά επίπεδα κοινωνικής προστασίας. Αυτός ο κοινωνικός πυλώνας αν θέλετε θα πρέπει να έχει τα μέσα έτσι ώστε να είναι αποδοτικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εκ νέου να καταστεί εν... μηχανή. η μηχανή για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και... Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ροντρίγκες. Ε, για την ECR θα λένε τον λόγο η κυρία Τρεμπέζιους παρακαλώ. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γιούνκερ. Δεν θέλω να είμαι αγενής, σίγουρα, αλλά είσαστε γέρος είσαστε κουρασμένος. Έχετε πλέον αναλώσει ό,τι μπορούσατε να αναλώσετε. Είσαστε εσείς υπεύθυνος για αυτή την Ευρώπη που αποτυγχάνει. Και τι κάνετε, επαναλαμβάνετε διαρκώς αυτές τις φράσεις ε, που λέγατε πάντα στο παρελθόν. Τίποτα καινούριο δεν μπορεί κανείς να αναμένει από εσά, αλλά από τη, παρά μόνο τη διαχείριση με κούραση αυτών όλων που είχατε διαχειριστεί κατά το παρελθόν και τα, που τα παρουσιάζετε εσείς σήμερα. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση Έχουμε και την ευρωκρίση και τις σοβαρές επιπτώσεις της. Έχουμε την ολέθρια ανεργία σε ε, υψηλότατα επίπεδα στη Νότια Ευρώπη. Έχουμε την κρίση μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην έχει ικανοποιητικέ απαντήσεις για αυτά τα προβλήματα. Λέτε ότι θέλετε καλύτερα να επεξηγήσετε λέει την πολιτική σας. Δεν χρειάζεται να την επεξηγήσετε κύριε Γιούγκερ. Πρέπει να είναι καλύτερη η πολιτική σας, να βελτιωθεί. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποτύχει στο μέλλον και να βρεθούν απαντήσεις για τα παιδιά μας για ένα μέλλον, καλύτερο μέλλον, ε, τότε σε σχέση με, τους, με τα όσα ο κύριος Φερχόφστατ είπε από τους αποκαλούμενους φιλελεύθερους, δεν είναι ο καλύτερος για να μας εκπροσωπήσει. Και σε σχέση με την, ε, τον ηγετικό ρόλο για το Brexit, είναι υπέρ του κεντρικού χαρακτήρα διαμόρφωσης της Ευρώπης και για την Ευρώπη à carte. Πιστεύω ότι η Ευρώπη à carte όπως αναφέρεται εδώ μπορεί να είναι η λύση για την Ευρώπη τώρα. Ευχαριστώ για την Ενωτική Αριστερά ο κύριος Φερέιρα τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Γιούγκερ. Εχθές ακριβώς η Business Europe, η Ένωση των Εργοδοτών, παρουσίασε τις παραγγελίες της ε, και το, το θεματολόγιο της. Ε, δεν πρέπει να είναι κανείς ε, ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τις συνόδους κορυφής, όπως συνέβη και με τη σύνοδο αυτή και τον λόγο που εκφωνήσατε. Αυτή είναι η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι άλλα για τους λαούς και τους πολίτες, για την ε, απασχόληση, για τους μισθούς, ε, για την κυριαρχία, για τα εργασιακά θέματα, με τις απειλές που διαμορφώνονται. Εδώ βλέπουμε τις κυρώσεις ε, που διαγράφονται κατά της Πορτογαλίας. Είπατε ότι είναι κατεπήγον. Ναι, αλλά είναι κατεπήγον να ξαναξεκινήσει η Ευρώπη. Η Goldman Sachs και τα Lux Leaks δεν θα είναι ποτέ η Ευρώπη των εργαζομένων και η Ευρώπη των λαών. Και αυτή είναι η κρυστάλλινη αλήθεια που είναι ομοί και πρέπει μια μέρα να το, να το δεχθείτε ότι θα εκραγεί κατά πρόσωπά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χότσον παρακαλώ στη συνέχεια. E η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια. Το δέχεται ο πρόεδρος Γιούγκερ αυτό. Και καλωσορίζω κάποιε από τι πρωτοβουλίε που ανέφερε, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει, όπω τη δημιουργία θέσεων απασχόλων, στη διασύνδεση και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πρόεδρο Γιούγκερ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη δύναμη στου πολίτε και να είναι αλληλέγγυα ο λαό τη Σκωτίας τον Ιούνιο ψήφισε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικοδομητικά να συνεργαστεί για να αντιμετωπιστούν οι συλλογικέ αυτέ απειλέ. Στην Σκωτία γίνονται προσπάθειε από όλα τα κόμματα για να δούμε ποια θα είναι η θέση τη Σκωτία, ιδίω ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Η κυβέρνησή μα ε, δουλεύει σκληρά για να πείσει την κυβέρνηση του Βασιλείου για να αναγνωρίσει τη δημοκρατική βούληση του λαού της Σκοτίας, όπως εκφράστηκε. Και ελπίζω η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα είναι ανοιχτό σε φάνταστες λύσεις, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ο δημοκρατικός ρόλος του σκοτσέζικου λαού. Σας ευχαριστούμε για την EFDD, η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εσείς επιβεβαιώσατε κύριε Γιούνκερ ότι λείπει στους πολίτες η Ευρώπη. Μιλήσατε για μια ιδανική Ευρώπη, μια Ευρώπη αλληλεγγύης, για μια Ευρώπη των πολιτών. και όμως το πρότυπο το οποίο προτείνεται δεν έχει σχέση με τις σημερινές ανάγκες. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αποτελεσματικές για τη διάσωση των τραπεζών, όχι όμως των προσφύγων και δεν μπόρεσαν να εγγυηθούν μια οικονομική ανάπτυξη για όλα τα κράτη-μέλη. Οι τεχνοκράτες, τα λόμπι, γενικά η ελίτ καθορίζουν τις διαδικασίες λήψεων αποφάσεων, επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, μειώνουν τη λαϊκή κυριαρχία, μειώνουν τη δημοκρατία, διαλύουν τις κοινωνικές κατακτήσεις, προωθούν τον υπερφιλελευθερισμό, την απορρίθμιση και οδηγούν στην φτώχεια και τις ανισότητες. Η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική πρόοδος των γενεών από το παρελθόν ε, δεν συνεχίζεται σήμερα και δεν αφήνουν τους πολίτες να γίνουν πρωταγωνιστές της μοίρας τους. Στη συνέχεια ο κύριος Σαλβίνη για την ομάδα INF. E ε, για μια ακόμη φορά ακούμε τις ίδιες αχλαμάρες. 3.000 νεκροί τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, εκατομμύρια ανέργων και παρόλα αυτά ποιοι είναι οι εχθροί της Ευρώπης, ε, οι εθνικιστές. Να πάτε σε γιατρό και σε έναν καλό γιατρό, αυτό σας χρειάζεται. Υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος για τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων. Αυτός ο κίνδυνος ε, είναι η Ισλαμική τρομοκρατία. Ε, κάθε βάρκα με πρόσφυγες που φτάνει στην Ιταλία τροφοδοτεί και σε χρήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό ε, τους τρομοκράτες στην Ευρώπη. Το εμπάργο στην ουσία οδήγησε σε απώλεια εκατομμυρίων από τους γεωργούς, δίδεται άχρηστα, ε, με άχρηστο λόγο θα έλεγα, χρήματα στην ε, ε, Τουρκία, καταπολεμάται την πολωνική κυβέρνηση, την οποία σέβομαι απολύτως, Νομίζω ότι είναι η τελευταία σας ομιλία σε αυτό εδώ το μέγαρο γιατί οι πολίτες δεν μπορούν και θέλουν πραγματικά λαϊκίστικα και εθνικιστικά να αφυπνιστούν πλέον. Θα λάβει το λόγο τώρα ο μη εγγεγραμμένος κύριε Ζόνεμπο, παρακαλώ. Ευχαριστώ αρχηγέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε. Όταν εγώ ανέλαβα την εντολή μου ήμουν υπέρ μια ισχυρής ε, Ευρώπης πυρήνα με 27 δορυφορικές χώρες. Τώρα μειώθηκε αυτός ο αριθμός μετά το Brexit ε, και μετά τα όσα συνέβησαν σε σχέση με την Ουγγαρία. Είμαι υπέρ του να δείξουμε την, την θύρα και στους Ιρλανδούς. Μια χώρα η οποία αρνείται να εισπράξει φόρους από μια εταιρεία όπως την Apple μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι μια Ευρώπη, θέλει μια Ευρώπη των επιχειρήσεων και όχι των πολιτών. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην Ιρλανδική κυβέρνηση Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ της Ιρλανδίας, αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι η Apple θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στην Ιρλανδία, ξεχάστε το η Apple μόνο ένα στόχο είχε, τη δημιουργία μιας θέσης απασχόλησης και αυτό απεβίωσε πλέον. Πάρτε λοιπόν αυτήν η σύστασή μου, πάρτε τα λεφτά και τρέξτε. Πρόκειται εδώ για δισεκατομμύρια. Θα δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες έτσι εσόδων για την ε, Ιρλανδία. Μπορείτε να αγοράσετε έτσι στο τέλος περισσότερα iPhones. Είναι μια κατάσταση ε, που θα είναι προς όφελος όλων με ένα ουισκάκι ξανασκεφτείτε τα. Παρακαλώ να πείτε σε σχέση με τον κύριο ε, Επίτροπο για τα επικοινωνιακά, ε, για αυτά τα θέματα για την προστασία στις Βρυξέλλες, την προστασία των καταναλωτών, να δράσει όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπορν για τον λόγο που εκφωνήσατε. Και επειδή με είπατε αρχηγό, αυτό με τιμά ιδιαίτερα που με αποκαλέσατε αρχηγό. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο αρχηγός ε, τέτοιου είδους ε, ε, ανθρώπων. Ευχαριστώ. Κύριε Λεβαντόφσκι, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σήμερα δεν είχαμε την ε, ε, συνήθεια αισιοδοξία όσον αφορά την κατάσταση της Ένωσης ε, διότι δεν ευσταθεί η αισιοδοξία δεν υπάρχει λόγος για αισιοδοξία και σε σχέση και με τον εορτασμό των συνθήκων της Ρώμης υπάρχουν πολλοί φόβοι και επιφυλάξεις και όλα αυτά παίζουν υπέρ των λαϊκιστών ξενοφοβία και λαϊκισμός επιβάλλουν προτεραιότητες και θεματολόγιο όσον αφορά τις συζητήσεις Υπάρχουν πολλές απειλές οι οποίες δυστυχώς τώρα είναι αυτές που συνενώνονται με τα φαινόμενα της μετανάστευσης και τα φαινόμενα της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν υπάρχουν κλωνοποιημένοι Νάιτζερ Φάρατζ σε πολλές χώρες ε, που δρούν προς την ίδια κατεύθυνση. Βλέπουμε τα θέματα τώρα της ασφάλειας εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης των συνόρων. Αυτή είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν αρχίσουν οι να σκέφτονται ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία θα εγγυηθούν την ασφάλεια, θα δίνουμε μια μάχη η οποία δεν μπορεί να κερδιθεί ποτέ. Θα είμαστε εμεί οι χαμένοι. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με τα όσα πρέπει να γίνουν δεν έχει κανένα νόημα να επικεντρωνόμαστε μόνο στην, πολυ... στην διαφορετικότητα. Πρέπει να αναζητηθεί ένας κοινό παρονομαστής. Αυτός δεν μπορεί να είναι ο ελάχιστος ε, κοινό παρονομαστής. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Έχει ζητηθεί παρέμβαση. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Εσείς μια και συζητάμε εδώ για τον λόγο του κυρίου ε, Γιούγκερ δεν έγινε αναφορά στα θέματα της οικογένειας και των δικαιωμάτων των οικογενειών. Οι οικογένειες βρίσκονται σε κρίση. Ποιοι είναι λοιπόν οι λαϊκιστές, γιατί φοβόσαστε να μιλήσετε για την οικογένεια, διότι αυτό θα οδηγούσε στην ανάληψη υποχρεώσεων απάντηση. Ο κύριος Γιούνκερ ο ίδιος επέλεξε το κείμενο το οποίο εξεφώνησε ως λόγο και νομίζω ήταν επαρκέστατος ο λόγος του. Μια επαρκέστατη απάντηση στη σημερινή κατάσταση. Ο κύριος Στάνισεφ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Πρόεδρε Γιούνκερ. Είχατε τη δύσκολη αποστολή να, οδηγη... να ηγηθείτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε... σε εποχές όπου το απίστευτο γίνεται πραγματικότητα. Το Brexit, η έλλειψη αλληλεγγύης για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των προσφύγων είναι απλώς τα συμπτώματα. Πώς θα βοηθήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια. Στα πέντε χρόνια της Επιτροπής ε, Μπαρόζο, η κοινωνική Ευρώπη έπεσε θύμα σε πολιτικές λιτότητας και μόνο. Όταν εσεί εκλεγήκατε ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποσχεθήκατε θα τα αλλάξετε αυτό. Είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τριπλό αλφα στα κοινωνικά. Αλλά δεν έχει γίνει πραγματικότητα αυτό. Και αυτό που περιμένουν οι σοσιαλιστέ από εσά και από την Κομισιόν είναι να έχετε ένα σαφέστατο δικό χάρτη, ο οποίο θα αντισταθμίσει την ε, ελεύθερη οικονομία και τι πρωτοβουλίε που σε αυτό το επίπεδο με σαφή κοινωνικά πρότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλώ ακόμα μια φορά να αντιμετωπίσετε σοβαρά το θέμα της νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικογένειά μας πρότεινε ένα σαφέστατο σχέδιο. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ε, νεολαία. Η απασχόληση με περισσότερα λεφτά από την εγγύηση για την νεολαία. Δεν άκουσα δέσμευση από εσά. Πολιτισμό, προστασία των παιδιών και εκπαίδευση. Εάν αρχίσετε τη μάχη για αυτά, υπέρ αυτών, τότε υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη να εξασφαλίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα λάβει τον λόγο στη συνέχεια για την ECR ο κύριος Τσίλε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σε ένα ιδανικό κόσμο καθένας θα αποκτήσει αυτά τα οποία επιθυμεί. Όλοι είναι κατά της λιτότητας, όλοι είναι υπέρ φυσικά της σωστής εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας αλλά νομίζω ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα. Εμείς τι κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικά μας. Εδώ βλέπω ότι οι ανισότητες αυξάνονται συνεχώς. Οι νέες γενιές της Ευρώπης την εγκαταλείπουν, προσπαθούν να πάνε αλλού. Εμένετε επίσης στην δημιουργία ενός νέου ταμείου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πώς θα το πετύχετε αυτό. Ε, είναι δυνατόν εμείς να προγραμματίσουμε τις δράσεις μας χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν είπατε τίποτα για τη Ρωσία. Είπατε ότι δώσατε αποζημιώσεις για τις απώλειες εισοδημάτων των γαλακτοπαραγωγών αλλά δεν είπατε τίποτα για την Κρυμαία, δεν είπατε για την επίθεση της Ρωσίας. Ένα λεπτό, η κυρία Ματίας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε λόγο για την κατάσταση της Ένωσης, αλλά συγκεκριμένα και να μην κάνουμε λόγο γενικόλογα η Γερμανία σε σχέση με τα δικά της πλεονάσματα όσον αφορά το παρελθόν αγνόησε και αύξησε τις επιδόσεις αυτές σε επίπεδα ρεκόρ αγνώντας το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και δεν τιμωρείται γιατί επειδή η Γερμανία είναι η Γερμανία η Γαλλία σε σχέση με τα όσα είχαν συμφωνηθεί παραβίασε το 2015 και εξακολουθεί να παραβιάζει το σύμφωνο αυτό και δεν τιμωρείται γιατί επειδή η Γαλλία είναι η Γαλλία. Και βλέπουμε εδώ ότι οι μεγαλύτερες και πιο επώδυνες προσαρμογές ε, που επιβλήθηκαν θα επιβληθούν τώρα κυρώσεις σε χώρες ε, που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό είναι πραγματικά επέσχυνο όταν συμβαίνει στην Πορτογαλία. Γιατί συμβαίνουν αυτά. Επειδή η Πορτογαλία είναι η Πορτογαλία. Αυτή είναι η κατάσταση της Ένωσης κύριοι. Και πείτε μου ένα πράγμα κύριε Πρόεδρε. Και εδώ δεν αισθάνεστε κάποια ντροπή. Δεν ε, υπάρχει κατεσχήνη για όλα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε για ένα λεπτό, Λούντγκρεν. Η Σας ευχαριστώ. Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ξέρουμε όλοι ποια είναι παρά τα όσα λέτε κύριε Γιούγκερ. Τα πράγματα εξελίσσονται ταχαίως και χάνεται η εμπιστοσύνη. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης ε, είναι αυτό που μας οδήγησε στο Brexit. Τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο Βρετανικός λαός μπορεί να απελευθερωθεί από, το, από την πότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Ενωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Ε, ο κύριος Γιούνκερ επίσης μίλησε για μια κοινή στρατιωτική ε, δύναμη και για μια κοινή άμυνα. Εμείς, ξέρετε, η χώρα μου ήταν πάντα μια ουδέτερη χώρα. Άρα θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η θέση μας αυτήν την ε, δύσκολη κρίση θα είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε σε μια τέτοια στρατιωτική συνεργασία. Επομένως, μπαίνει αυτό το θέμα της ε, εμπιστοσύνης ακόμα πιο επιτακτικά και στο μυαλό των ψηφοφόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένας ε, μεγάλος ασθενής, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ο κύριος Φιλίπς, για ένα λεπτό, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ίδια, με το άτομο του Προέδρου της ε, αναφέρεται σε υπαρξιακή κατάσταση, υπαρξιακή κρίση. Είναι ολέθρια η κατάσταση. Οι Βρετανοί καλά είπαν θα εγκαταλείψουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ή την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει καταδίκη της Πολωνίας με πλειοψηφική απόφαση και από το Λουξεμβούργο ζητείται τώρα ο αποκλεισμό ε, της Ουγγαρίας. Πόσο παράλογα μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Δεν αλλάζει δηλαδή τίποτα αντί αυτά τα ζητήματα ζητήματα να μπορέσουν να διαμορφωθούν και να επιληθούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας ε, για την ανάπτυξη ώστε να υπάρξουν θετικές προοπτικές. Αλλάζουν τα πράγματα και εδώ πραγματικά υπάρχει μια πολύ αρνητική ε, τροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ενιαίο νόμισμα και όσον αφορά τις ε, σημερινές εξελίξεις. Κατανοήστε επιτέλους τις εξελίξεις όσον αφορά το δημοψήφισμα των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Βρετανία επιστρέψουμε στο κράτος δικαίου, στην επικουρικότητα, στα κυριαρχικά δικαιώματα και τότε θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορητής για 1,5 λεπτό, Λαμασούρ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτέλους, τα πρώτα θεμέλια μιας ε, Ευρώπης άμυνας ε, τα διαβλέπουμε, χαιρόμαστε. Αλλά μην ξεχνάμε Όπω σωστά υπενθυμίσατε κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή ότι τα στρατιωτικά μέσα είναι ένα απλό εργαλείο στην υπηρεσία μια εξωτερική πολιτική. Πολύ σωστά, δώσατε το παράδειγμα τη Συρίας. Εγώ θα αναφέρω δύο άλλα. Ποια είναι η εξωτερική μα πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Η συμφωνία του Μίσκ δεν την διαπραγματεύτηκε η Ένωση, αλλά δύο κράτη-μέλη. Και πέρα από την Ουκρανία, η κατάσταση στον Κάφκασο, οι απειλέ στι στις χώρε. Η διπλωματία για το φυσικό αέριο της Ρωσίας είναι ουσιαστικά θέματα που τα αγνοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απίθανο που 25 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου είμαστε ανίκανοι να μιλήσουμε με μία φωνή απέναντι στη Μόσχα. Δεύτερο παράδειγμα, Λιβύη. Ξανά γίνε η πρώτη πύλη εισόδου ε, μεταναστών και κυκλοφορούν οι τρομοκρατικές ε, ισλαμικές ε, πολιτοφυλακές. Κατάρ, ε, Τουρκία, Αίγυπτος. Κάνουν κάποιες συμφωνίες με κάποια κράτη-μέλη. Πού είναι η Ευρώπη? Στη θάλασσα. Στα ανοιχτά, στο πέλαγος. Για ανθρωπιστικές βοήθειες, σίγουρα. Αλλά όμως αναγκάζεται να υφίσταται αποφάσεις που παίρνουν άλλοι. Χωρίς κοινή πολιτική εξωτερική θα έχουμε επιπλέον μέσα για να συνεχίζουμε να μην κάνουμε τίποτα μαζί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό ο κύριος Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Μία πτυχή μόνο από τον λόγο του κύριου Γιούγκερ θα επιλέξω και θα αναφερθώ σε αυτήν. Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια. Ασφάλεια εσωτερική και ασφάλεια εξωτερική. Και γι' αυτό κύριε Γιούγκερ σας υποστηρίζω απόλυτα για τις προτάσεις σας για την καλύτερη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών. Επίση, υποστήριξη για ένα ταμείο για την πολιτική άμυνα. Επίση, όσον αφορά την προώθηση τη διαρθρωμένη δομημένη συνεργασία σε αυτού του τομεί. Αλλά όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και όχι σε έναν παράλογο επιπλέον εξοπλισμό. Και γι' αυτό αυτέ οι δραστηριότητε που επιθυμούμε μόνο τότε μπορούν να είναι λειτουργικέ και αποτελεσματικέ όταν θα είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να διαθέσουν πρόσθετα κονδύλια για τέτοιου είδου πρόσθετε χρήσει. Η ασφάλεια των εξωτερικών σύνορων μα. Ο έλεγχο να ξέρουμε ποιοι περνάνε τα σύνορα αυτά μπαίνοντα και βγαίνοντα. Ναι, έχουμε αμελήσει αυτή την πτυχή. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα γι' αυτό. Ένα όμω πρέπει να είναι σαφέ. Δεν είναι αυτή η λύση για τα προβλήματα τα μεταναστευτικά και την κρίση προσφύγων. Το πολύ πολύ σε σχέση με την κατανομή προσφύγων ίσω θα βοηθήσει να απαμπληθεί, να ανακουφιστεί. Η, η κρίση των προσφύγων θα επιληθεί μόνο όταν οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ληφθούν σοβαρά από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τα αίτια των διωγμών και της φυγής αυτών των προσφύγων από τις χώρες τους αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. For one and a half minutes, Mr. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Γκονθάλεθ Πόνς. Κύριε Γιούγκερ, η Ευρώπη είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Οι απόπειρες οι εγκληματικές, τα τρομοκρατικά πλήγματα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, όλα όσα έχουν γίνει αναδεικνύουν και αναπτύσσουν τον λαϊκισμό και την ξενοφοβία. Την εντύπωση ότι το σύστημα δεν λειτουργεί. Τα θεσμικά όργανα λειτουργούν. Λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν λειτουργεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών. Χωρί αλληλεγγύη δεν θα μπορέσει να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και όταν λειτουργούν τα θεσμικά όργανα. Αλληλεγγύη είναι αυτό που μάθαμε από του πολέμου αλληλεγγύη είναι όπως είπατε κύριε Γιούγκερ, κύριε Βέμπερ, ένας τρόπος ζωής των Ευρωπαίων. Τρόπος ζωής που θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών, όχι υπέρ κάποιων και λιγότερο για κάποιους άλλους. Όταν τα κράτη θα υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους ε, για τους προϋπολογισμούς, ε, αλλά επίσης ε, αλληλεγγύη όταν οι εταίροι δεν θα αναζητούν να επιβάλλουν κυρώσεις εις βάρος άλλων. Αλληλεγγύη είναι να κατανοήσουμε ότι η μαζική μετανάστευση είναι κοινό πρόβλημα όλων. Αλληλεγγύη είναι μια ενιαία οικονομία για όλα τα κράτη-μέλη και όχι 28 ξεχωριστέ οικονομίε. Αλληλεγγύη είναι 27 κράτη υπέρ ενό, ένα υπέρ όλων των 27. Αυτό είναι το εφικτό και δυνατό για τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό σας δίνω συγχαρητήρια για το λόγο που εκφωνήσατε. Βασιστείτε στη δική μου υποστήριξη και την υποστήριξη τη χώρα μου της Ισπανίας. Τώρα για ένα λεπτό κυρία παρακαλώ. Uh, Υπάρχει όμως μπλε κάρτα από συνάδελφο πρώτα. Για σας κύριε Γκοθάλετ Πόνς, την δέχεστε. Λοιπόν, παρακαλώ για την ερώτησή σας. Έχετε τον λόγο συνάδελφε. Ε, ε σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πόνς, εσείς θεωρείτε ότι είναι δίκαιο η Ισπανική κυβέρνηση να προαναγγέλει περισσότερα μέτρα περικοπών για το επόμενο έτος 2017 για να συμμορφωθεί με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα θα πλήξουν ιδιαίτερα εκείνους που είναι σε πιο μειονεκτική θέση στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόνς για να απαντήσει. Πιστεύω ότι η Ισπανία όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Αν είμαστε μια ενιαία οικονομία πρέπει να φερόμαστε με νομιμότητα και με θεμητό τρόπο νόμιμα σε σχέση με τους άλλους. Δεν πιστεύω ότι θα υποστεί κυρώσεις η Ισπανία, αλλά πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων η Ισπανία και να τηρεί τα υπεσχημένα. Το να τηρεί κανείς τον λόγο που έδωσε είναι ένδειξη καλού εταίρου. Τώρα η κυρία Φαζό. Στάνιε. Πρόεδρε, η δυσπιστία είναι αυτή που βασιλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί Ευρωπαίοι έχουν ξεχάσει και την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Δεν το ξέραν ποτέ, δεν το μάθαν ποτέ. Γιατί, Γιατί πάρα πολλοί πολιτικοί ξέχασαν τις ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί δεν αποφασίσ... με αποφασιστικότητα αντιδράσαμε στην παραβίαση των δικαιωμάτων μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν προσφέρουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Η μακροπρόθεσμη, ε, το μακροπρόθεσμο όραμά μας θα πρέπει να βασιστεί σε αλληλεγγύη και όχι σε μυστικές συμφωνίες. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε την ασφάλεια και παράλληλα να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει οι πολίτες να προστατεύεται η ιδιωτική του σφαίρα. Κύριε Γιούγκερ Καλό είναι οι νέοι, με αυτά που είπατε, να βοηθηθούν και να ενταχθούν. Αλλά χρειαζόμαστε αισιοδοξία, γιατί η απεσιοδοξία δεν λύνει τα προβλήματα. Και όλοι όσοι από εμά έχουν υπεύθυνε θέσει και αξιώματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επόμενοι μήνε είναι κρίσιμοι. Που θα μετρήσουν αν η Ευρώπη θέλει να αντισταθεί στο λαϊκισμό. Ο κ. Τσέδα, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η παρέμβασή σας ήταν ξεκάθαρη σε αυτή την κρίσιμη και ιστορική στιγμή. Τα λόγια σα μα κάνουν να διαβλέπουμε ένα φω στο βάθο του τούνελ μετά από μια μακρά κρίση. Βλέπουμε όμω ένα ξερό όχι ε, απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα από ένα πολύ σημαντικό κράτο. Και περιμένουμε ευθύνη και υπευθυνότητα από αυτό το κράτο και πρέπει να δείξουμε και εμεί υπευθυνότητα. Κάθε μέρα βλέπουμε να αυξάνει η δυσπιστία των πολιτών μα απέναντι στην Ευρώπη. Όπω ε, είπατε κι εσεί, Ζητάμε από την Κομισιόν ε, ένα ποιοτικό άλμα. Πρέπει να δείξουμε φιλοδοξία και συγκεκριμένου στόχου. Θα πρέπει να υπάρξει ασφάλεια, ε, να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση, να, υπάρξει, ε, να υπάρξουν θέσει απασχόληση και προστασία τη αποταμίευση. Για την ασφάλεια θα πρέπει να έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Αστομία Συνόρων, πρέπει να ενισχυθεί, αλλά χρειαζόμαστε ένα πραγματικό στρατό και μια κοινή εξωτερική πολιτική. Είναι απαραίτητο αυτό για να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ειρήνη μας για πολλά χρόνια, που είναι το αποτέλεσμα 60 ετών κοινή ύπαρξη. Η ανεργία, κυρίω των νέων στην Ευρώπη, ξεπέρασε το 20% και στη χώρα μου φτάνει στο 40%. Το σχέδιο των επενδύσεων δίνει τα πρώτα αποτελέσματα. Καλό είναι που θα το ενισχύσετε, μακάρι να τριπλασιάσουμε τους πόρους. Ας ε, τονίσουμε τις ε, επενδύσεις, ούτως ώστε να υπάρξει και ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Η προστασία των καταθέσεων πρέπει να εξασφαλιστεί. Πιστεύουμε ότι με ιδιωτικού πόρου θα έπρεπε κανονικά να προστατεύσει τους ε, πολίτες. Μπορεί να του προστατεύσει όμως. Γιατί νόμιζα ότι προστατεύεται μόνο τον ε, προπολογισμό των κρατών. Στην Ευρώπη, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη απόκριση. Είναι και η ώρα, κύριε Γιούγκερ, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με δύναμη και αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι θέλετε να ακούσετε θετικές προτάσεις. Ε, πολύ σωστό αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα μετά το Brexit να πέσουν όλοι σε μαζική κατάθλιψη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες συνθήκες ε, και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση με θετικό τρόπο. Σίγουρα οι πολιτικές ομάδες ε, θα πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσουν να καταλήξουν σε λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως της ανεργίας των νέων και θα πρέπει να ε, αποδώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, διότι μην ξεχνάμε ότι οι νέοι επιθυμούν μια διαφορετική Ευρώπη. Επιμείνατε και εσείς σε σχετικές πρωτοβουλίες. Ε, λοιπόν, ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα βιομηχανία, μια μετάβαση σε νέα κατάσταση. Οι επενδύσεις ε, θα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτή την μετάβαση. Ευχαριστούμε κύριο Σάιρ. Μιλήσατε με κατηγορηματικότητα για την ασφάλεια το ΕΛΚ χαιρετίζει το γεγονός ότι στον τομέα της ασφάλειας ε, έχει πλέον ε, δικό του επίτροπο και πρέπει να προχωρήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνω λοιπόν το Κοινοβούλιο να έχει μια μόνιμη επιτροπή για την εσωτερική ασφάλεια. Έχουμε τα περίπλοκα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας και τα θέματα αυτά αποτελούν μία μόνο διάσταση στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ ομιλώ για την κρίση μετανάστευσης ως πολιτικός. Η δική μας η θέση είναι σαφής και ανθρώπινη. Αντί δηλαδή να μεταφέρουμε τα προβλήματα στην Ευρώπη, καλύτερα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται ε, η βοήθεια να τους δίδεται έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να συγκρατηθεί η παράτυπη μετανάστευση. Ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη της γης ε, μπορούν να έρχονται στην Ευρώπη και να ε, καταεπιμερίζονται με ε, κάποια κλίδα. Οι Ούγγροι θα αποφασίσουν στις αρχές του Οκτωβρίου και θα αποφασίσουν ειλικρινά. Έχετε μία ερώτηση από τον κύριο Ιουτσέτσι. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα δημιουργηθεί το ανώτατο όριο. Ο συνάδελφος κύριος Φίντες μίλησε για ανθρωπιά και πώς μπορεί να κοιτάει τον κύριο Γιούνκερ στα μάτια τη στιγμή που στην Ουγγαρία γίνεται εκστρατεία με δημόσια κονδύλια και όπου στην αφή αυτή βλέπουμε το πρόσωπο του κυρίου Γιούγκα ε, στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ σαν ένα είναι ο κύριος Γιούγκερ υπεύθυνο για το ότι υπήρξε τρομοκρατική επίθεση στο Ζάβεντεμ και εσείς μιλάτε για ανθρωπιά ε, λυπάμαι πάρα πολύ ε, ξεπεράσετε το χρόνο σας τέλος πάντων έχετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση κύριε πρόεδρε ερώτηση δεν άκουσα ωραία Περνάμε στον επόμενο μιλητή για ένα λεπτό, η κυρία Τόμας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα ποιητή ε, Γαλλό που λέει ότι δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχουν μόνο αποδείξεις αγάπης. Ε, η δήλωση αγάπης που κάνετε στην Ευρώπη δεν φτάνει λοιπόν, χρειάζονται αποδείξεις. Πόσα χρόνια περιμένουν οι πολίτες το κοινωνικό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει ότι δεν το πιστεύουν πλέον και 80% της νομοθεσίας ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν έχουμε αποδείξεις έδρακτες ε, της δέσμευσής μας μέσα στο προϋπολογισμό. Γι' αυτό έχουν ακινητοποιηθεί τόσες οι διαδικασίες. Θα πρέπει να περάσουμε στο έργο, θα πρέπει να εξισώσουμε τις πολιτικές μας δηλώσεις με συγκεκριμένες δράσεις, ξεκινώντας με πραγματική αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και του προϋπολογισμού μας για το 2017, κάθε νέα πολιτική απόφαση, σαν αυτή που ανακοινώσατε σήμερα και που μας βρίσκει σύμφωνους ε, για τα σύνορα, για την άμυνα, θα πρέπει να συνοδεύεται από οικονομικούς πόρους. Όμως ε, δεν πρέπει να πούμε όχι στις περικοπές για την έρευνα, δηλαδή ε, είναι οι επενδύσεις που θα κάνουμε στο μέλλον. Ε, η εγγύηση για την νεολαία που αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε αναλάβει καμία δέσμευση για τον προπολογισμό του 2017. Η κυρία Τόμα, τελευταία πρόταση. Πρόεδρε και Προεδρεύοντα το Συμβούλιο, περιμένουμε αυτή την πρωτοβουλία, τόσο ώστε να έχουμε νέους ίδιους πόρους. Περιμένουμε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπραγμάτευση με όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ε, ο... Φυσικά θα πρέπει να δείχνει ευελιξία ο Πρόεδρος, όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου και την, ε, το χρόνο. Ο κύριος Δρανζέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ομιλία σας. Είναι ε, σημαντικότατα, σημαίνει προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλήσατε για συγκεκριμένα μέτρα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να θέσουμε το εξής ερώτημα όμως. Μας ανησυχεί ο λαϊκισμός ε, ευρωσκεπτικισμός. Όμως, τι βλέπουμε ε, στα προπήρια των ευρωπαϊκών θεσμών για τη δυνατότητα, ε, το ενδεχόμενο περικοπής ε, των ε, κονδυλίων των διαρθρωτικών τεμένων για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Μα έκαναν πελώριες θυσίες ή προτίθενται να υλοποιήσουν τα μέτρα. Δεν πρέπει να τους μεταχειρίζεστε έτσι. Το κράτος ε, της Πορτογαλίας. Ε, μην ξεχνάτε, ο λαός της Πορτογαλίας, ε, οι εταιρείε, οι πολίτες, τα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να τιμωρούνται μέσα από την στολή χρηματοδότησης. Και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία ο καλπάζων λαϊκισμός είναι που αντιβαίνει στο σχέδιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Χόλτσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν είναι λόγο για να επιχαίρουν ορισμένοι. Και μερικοί το πράττουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Εμεί δεν εκλεγήκαμε για να είμαστε ε, καταστροφικοί, αλλά εκλεγήκαμε για να αντιμετωπίζουμε τι δυσκολίε ω πρόκληση. Και η Ευρώπη ανέκαθεν ε, προχωρούσε και πρόοδευε οποτεδήποτε επίλυε τις δυσκολίες τη. Αλλά δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, στο προσφυγικό, στη θεσμική κρίση, στην οικονομική κρίση. Να μην περιοριζόμαστε βέβαια μόνο σε αυτά, αλλά να στρέφουμε το βλέμμα και προ το μέλλον. Και το βρίσκω ιδιαίτερα θετικό, κύριε Γιούγκερ, το ότι δίδεται ιδιαίτερο περιθώριο στην ευρυζωνικότητα. Η ψηφιακή πρόοδο είναι σημαντική, η ψηφιακή αγορά είναι το σημαντικότερο εγχείρημά μα, γιατί είναι εκείνο που διασφαλίζει τι θέσει εργασία. Και όσον αφορά και το πακέτο προστασία δεδομένων, διαπιστώσαμε ότι εμεί ω Ευρωπαίοι μπορούμε να καθορίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις προδιαγραφές. Ο κύριος Κάρας, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κυρία ε, Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε Γιούγκα, με την παρουσίαση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης που παρουσιάσατε, μας ικανοποίησατε γιατί απαριθμίσατε και ονοματίσατε τις προτεραιότητες. Το θέμα είναι πώς ορισμένοι πολιτικοί θα αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, τις ανησυχίες των ανθρώπων, ε, τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μερικές φορές ε, Ορισμένα κράτη δηλιάζουν και δεν λένε την αλήθεια στους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν ας αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αντί να αφήσουμε να μας γονατίσουν. Ο λαϊκισμός ε, ε, οδηγεί σε υποχώρηση, οπισθοχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πρατισλάβα θα πρέπει να έχουμε ένα μήνυμα ε, της αλληλεγγύης, να υπάρξει μια αντιστροφή. Τώρα πλέον πρέπει να προχωρήσουν όλα μαζί τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια για περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη, για τον διπλασιασμό του προγράμματο επενδύσεων, για την ψηφική αγορά, για την κατανομή των προσφύγων, επίση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και για την κοινή πολιτική μετανάστευση και χορήγηση ασύλου. Ο κύριο Κόρμπετ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Το Brexit είναι ένα από αυτά μόνο. Ε, αποτελεί την ε, μητέρα όλων των διαζυγίων και αν γίνει πρόχειρα θα αποτελέσει καταστροφή και για τις δύο πλευρές. Τα συζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν είναι πάρα πολλά και κάθε μέρα ανακαλύπτουν και καινούρια τα οποία ποτέ δεν είχε αντιληφθεί και δεν είχε σχολιάσει η εκστρατεία υπέρ του Brexit. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 50 ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχει σαφή ιδέα για το τι θέλει να κάνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Το μεγαλύτερο από, αυτό, από αυτά είναι το κατά πόσον η Βρετανία θέλει να διατηρήσει τη θέση της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αν όμως είναι έτσι, πράγματι θα πρέπει να δεχτεί και όλους τους κανόνες της ενιαίας ε, αγοράς. Αν θέλει να την εγκαταλείψει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει καινούριου φραγμούς στο εμπόριό της, δασμολογικούς και άλλους οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην ε, Βρετανία και στην Ευρώπη. Αυτοί όμως που ψήφισαν υπέρ του Brexit λένε πλέον και παραπονούνται ότι δεν ψήφισαν για αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πολλοί ζητούν να το ξανασκεφτούν. Ευχαριστώ πολύ. Μπλε κάρτα από τον κύριο Σμιτ. Τη δέχεστε, κύριε Κόρμπετ. Ναι. 30 δευτερόλεπτα. Ε, χαίρομαι που ο κύριος ε, Κόρμπετ ε, επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για το ευρωπαϊκό πνεύμα θα συμφωνούσατε κύριε Κόρμπετ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια κοινή αντίληψη μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά την έξοδο του Βασίλειου από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα περιλαμβάνει το Γιβλαρτάρ, τη Σκωτία, την Βόρεια Ιρλανδία κλπ. Και ότι θα πρέπει η πολυφωνία μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλιστεί με ευελιξία και να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση που θα παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Yes, I agree. Απάντηση. Ναι, η κατάσταση αυτή δημιουργήσε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ποτέ δεν τα είχαμε συζητήσει πριν λάβουμε την απόφασή μας και σίγουρα κανείς δεν, από αυτούς που θέλαν να βγάλουν την Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα είχε θίξει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλα τα τμήματα της Βρετανίας προκειμένου να βρούμε μια λύση. Και όταν κάποια στιγμή ο λαός καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα και πόσο διαφέρει από τις υποσχέσεις και τα ωραία λόγια που είχαν λεχθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, τότε πολλοί Βρετανοί πιστεύω ότι θα πούν θέλουμε να το ξανασκεφτούμε. Σουίτσα. Κυρία Σουίτσα, ένα λεπτό. Ναι, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παραφράσω τον κύριο Μάνφρετ Βέμπερ που είπε πρέπει, ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το λαϊκισμό εναντίον των Βρυξελών. Ε, η δική μας υποχρέωση ε, είναι να δίνουμε θετική σκέψη και θετικά επιχείρηματα για την Ευρωπαϊκή και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Γιούνκερ. Έτσι όπως μίλησε θα πρέπει να μιλάμε και εμείς στα εθνικά μας κοινοβούλια. Είναι αλήθεια ότι έχει διαβρωθεί μετά τον Brexit κατά κάποιο τρόπο η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απομονωθεί, δεν μπορεί να εργαστεί από μόνη της και τα προβλήματά της δεν είναι δυνατόν να επιληθούν μόνο στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Πρέπει να επιληθούν και στην Αθήνα και στη Μαδρίτη και στο Ζάγκρεπ. Ο κύριος Πλάνκοβιτς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος ε, ο Πρωθυπουργό τη ε, Κροατία και είμαι σίγουρο ότι θα συνεισφέρει στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γιούγκερ, σα ε, βεβαιώνω ότι θα σα βοηθήσουμε στην επίτευξη των κοινών μα στόχων. Θα ήθελα τέλο να σα ευχαριστήσω που εργάζεστε έτσι ώστε οι εργαζόμενοι όπου και να βρίσκονται θα έχουν τον ίδιο μισθό και τα ίδια δικαιώματα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο σεβόμαστε την αρχή της ελεγγύης Ευρωπαϊκής ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Τόγια, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ε, που πρωταγωνιστούμε σήμερα στην Ευρώπη σίγουρα δεν είμαστε ήρωες και ίσως ε, τα καθήκοντα και υποχρεώσει να μας ξεπερνούν και από τις ε, δικές μας τις επιλογές προκύπτουν ιστορικές αποφάσεις. Θα αξιολογηθεί η Ευρώπη πώ αντιμετώπισε μια σημαντική κρίση, κατά πόσον κατόρθωσε να αναγεννηθεί ή να διαλυθεί. Ο κυριο Γιούγκερ πολύ σωστά μα τα επενθύμισε όλα αυτά. Η δική μας ευθύνη σήμερα δεν συνδυάζεται με την καθημερινή μας πολιτική ζωή μας συνδυάζεται ακριβώς με αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Άρα δεν λέμε ναι, ίσα, λέμε όχι σε οποιασδήποτε ε, αρνητικές στάσεις. Ε, εμείς θεωρούμε ότι ε, πρέπει να αναστηθούν νέε πολιτικές και στο Brexit. Να ξεκινήσουμε μια νέα πολιτική, το τέλος θα πρέπει να είναι μια πραγματική επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα επίσης να πω ότι όπως και άλλοι θα πρέπει οι συνθήκες να εφαρμοστούν με ευφύη τρόπο και να μην χάσουμε την αξιοπιστία μας γιατί αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο εναντί των πολιτών και θα πω δύο πράγματα ισοτιμία και δικαιοσύνη φορολογική αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής υπάρχει μία πρόταση αυτή η ασφάλεια για τους άνεργους. Αυτό πρέπει να ενταχθεί στην κοινωνική πολιτική της Ευρώπης για να δείξουμε ότι εμείς και πιστεύω ότι και εσείς το πιστεύετε για να αποδείξουμε λοιπόν ότι εμείς πραγματικά αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια των αδύνατων πολυσυμπολιτών μας. Είναι πρόταση πάντων. Γι' αυτό λοιπόν ας το κάνουμε αυτό την αυαρχίδα της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Ο κύριος Μπούλμαν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, πολύ σωστά είπατε ότι πάρα πολλά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν εξελίσσονται όπως θα έπρεπε και σε πάρα πολλούς τομείς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη αλληλεγγύη. Ακόμα λοιπόν ε, και αν εμείς ε, λέμε ότι θα πρέπει να δείξετε θάρρος, να προχωρήσετε, να δώσετε τον τόνο για μια θαραλέα ειλικρινή Ευρώπη, ξέρουμε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε εύκολα. Πάρα πολλά πράγματα πράγματα γίνονται μόνο ε, σε εθνικό επίπεδο. Μιλάτε για ευθύ κανόνε και θα πω κάτι, μια πρόταση που την καταθέσαμε πριν από πέντε χρόνια στο πλαίσιο τη συζήτηση για το Σύμφωνο Σταθερότητα. Θα πρέπει να είναι τελείω διαφορετικό το κατά πόσον μια χώρα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ανεργία ή κατά πόσον διατηρεί τον υδροκεφαλισμό στην διοίκηση. Θα πρέπει να κάνει διαφορά κατά πόσον μια χώρα επενδύει στην ενεργειακή αλλαγή ή θέλει να επανέλθει στην παλαιολιτική εποχή. Είναι διαφορετικό το αν μια χώρα βοηθάει με αλληλεγγύη τους πρόσφυγες και τους προσφέρει νέες αιστείες ή το κατά πόσον δεν τους τίνει καμία χείρα βοηθείας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει ένα ανεξάντλητο δυναμικό για δημιουργικότητα. Οφείλουμε να αλλάξουμε τους δημοσιονομικούς μας κανόνες έτσι ώστε και η Κομισιόν να είναι ευφύης στην καθοδήγησή της. Αυτό είναι το έτοιμά μας και περιμένουμε τις προτάσεις σας. Για ένα λεπτό, κυρία Γκαρσία Περές. Ε, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνονται, εθνικισμοί διευρύνονται μεγαλών. Αυτό είναι η σύνοψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Όμως είναι στα χέρια μας να το αλλάξουμε. Με μια κοινή προσπάθεια μπορούμε να σώσουμε το ευρωπαϊκό ε, όραμα γιατί οι διάφορες κρίσεις, η οικονομική, η προσφυγική κλπ. έχουν μόνο κοινέ λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Γιούνκερ ως επικεφαλής ε, θα πρέπει ε, να αντιταχθούν σε αυτούς που μπλοκάρουν τις ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες. Θέλουμε να δείξει μεγαλύτερη επιμονή. Θέλουμε μια πιο δίκαιη δημοσιονομική πολιτική δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Ε, δεν θα πρέπει να μπλοκαριστούν οι, τα κονδύλια για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα το κάνουμε συνεργαζόμενοι, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να χαθεί η ελπίδα για το ευρωπαϊκό όραμα. Δεν θα επιτρέψουμε να χάσουμε την πίστη μας στο ότι είναι δυνατή μια καλύτερη Ευρώπη. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων ζητούν το λόγο. Εσείς θέλετε το λόγο κυρία μου ή έχετε μπλε κάρτα. Μπλε κάρτα. Α, catch the Ωραία. Σας προσθέτουμε και εσάς τον κατάλογο. Ο λόγος στον κύριο Κιώτος. Για ένα λεπτό και θα είμαι πολύ αυστηρή. ναι, εσείς είσαστε, παρακαλώ. Δεν ήθελα να σας πω, κύριο, τη θέση 584. Ζητώ συγγνώμη παρέστηρα το όνομά σας. Για να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εγώ προτείνω δύο. Πρώτον, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία, την οποία θεωρώ σημαντική χώρα με την οποία πρέπει να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας, αλλά δεν μπορεί να θεωρούμε ότι η Τουρκία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο αφήνουμε την εκκρεμότητα να αιωρείται, τόσο θα δημιουργείται δυναμική τύπου Brexit και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούν αδιανόητη την προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας χώρας με τόσα αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε σε σημαντική αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τον οποίο δυστυχώς μειώνουμε τα τελευταία χρόνια, για να χρηματοδοτήσουμε την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, την έρευνα, την καινοτομία και ένα σημαντικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα υπέρ της απασχόλησης των νέων. Πιστεύω ότι μπορούμε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν πραγματικά θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κίρτσο. Για ένα λεπτό. Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γιούγκερ, το είπατε κι εσεί. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση σήμερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Από όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για την κατάσταση της ε, Ένωσης ε, Προεδρίας ε, Μπαρόσο, δεν είδαμε χειρότερο σύμπτωμα της χειροτέρευση κατάστασης από το Brexit και την απόσταση μεταξύ ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. Η, τα δικά σας ε, λόγια ε, είναι πραγματικά πολύ όμορφα, αλλά οι πράξεις σας έχουν μείνει πίσω, υστερούν. Ε, η ανάπτυξη είναι ελάχιστη. Βλέπετε ότι το πρόγραμμα Juncker δεν αρκεί. Η ανεργία των νέων, ψηλότατη υψηλότατη, δεν λειτουργεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ε, έχουμε τις απειλές για πρόστιμα στην Ισπανία και την Πορτογαλία που έχουν κάνει τόσο πολλές προσπάθειες και παρόλα αυτά δέχονται απειλές. Και βέβαια έχουμε και το θέμα της απειλή σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για την αποδοχή των προσφύγων. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ιδεών, αλλά έλλειψη πολιτικής ε, βούλησης ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank Φαντάζομαι ότι έχετε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το ρολόι. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, αν δεν στο μεταξύ δεν φτιαχτεί. Ένα λεπτό παρακαλώ να τηρείτε ο χρόνος. Φόρντ. Ε, ε, κύριε Γιούγκερ, αναφερθήκατε στο, στα κηρύγματα και στα εγκλήματα μίσους. Έξι ε, ε, συλλήψεις είχαμε την περασμένη εβδομάδα, όμως γιατί δεν αναφερθήκατε στις ε, ε, εκατοντάδες ανθρώπων στο Έσεξ που σύσσωμε καταδικάζουν τη δολοφονία αυτή και η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών επιθυμούν ειρηνικές ε, ε, διαπραγματεύσεις για το Brexit. Υπάρχουν βαθύτατοι εμπορικοί δεσμοί ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ξεριζώσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο από την εσωτερική αγορά χωρίς μακροπρόθεσμο προγραμματισμό θα υπάρξουν κοινωνικέ επιπτώσει που θα πλήξουν ολόκληρη την Ευρώπη. Αμφωτέρων των πλευρών οι διαπραγματευτέ θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο σε αυτέ τι διαπραγματεύσει ε, για να έχουν σωστά αποτελέσματα. Ε, κυρία Γεωργίευα, θα ήσασταν καταπληκτικοί σε μια θέση στον ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Μας τουπλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ε, πρέπει να ασκήσουμε αυτοκριτική. Δεν υπάρχουν πραγματικά μέτρα ε, για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Είναι πολλές οι κρίσεις, κρίσεις που εξελίσσονται παράλληλα. Και αυτό λοιπόν ε, φαίνεται από το ότι οι λύσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι αναποτελεσματικές. Οι περισσότεροι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου βλέπουν ότι το μέλλον τους δεν είναι η Ευρώπη. Υπάρχει και κρίση ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο. Καμία κρίση δεν είναι μοιραία, όμως κρίσεις οφείλουν να μας οδηγήσουν στο να κατανοήσουμε το αίτιο και το αιτιατό. Ε, να αποδώσουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι και να ονοματίζουμε τους ανθρώπους, να πούμε ποιοι εν πάση περιπτώσει έκαναν τα λάθη. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει πραγματικά να λάβει υπόψη του κατά πόσο μπορεί να οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός κρίσης ή αλλιώς να παραιτηθεί. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση της Ένωσης είναι ανάλογη. Πριν από δύο χρόνια ε, σας ψήφισα γιατί μας ε, υποσχεθήκατε τότε ότι θα κάνετε μεταρρυθμίσεις που θα καταργήσουν τα εθνικά σύνορα. Θα ε, κινητοποιούσατε το ψηφιακό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν όλα πιο εύκολο να γίνουν κατανοητά. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή ούτε καν σχεδόν να θίγετε τα θέματα του copyright που είχατε υποσχεθεί παλαιότερα θα το κάνετε και ανταυτού λέτε ότι οι εκδότες ε, πρέπει να πληρώνονται για τα link που οδηγούν στα άρθρα τους. Ε, το θέμα είναι ότι είναι πλέον πλέον πιο δύσκολο για τις ε, τεχνικές εταιρείες ε, να ανταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε λιγότερα link σε ευρωπαϊκές δημοσιεύσεις και σε τελική ανάλυση η πρόταση αυτή έχει απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολλές φορές. Ένα λεπτό, επιτίδιος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τα όσα μας ανέφερε ο κύριος Γιούγκερ στην ομιλία του δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια επανάληψη γνωστών ήδη αναλύσεων ε, φιλολογικού περιεχομένου ε, θέσεων και ανεφάρμοστων επιδιώξεων. Πώς είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να γίνει η επανένωση της Κύπρου όταν η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται αυτή την κατάσταση πώ είναι εδώ να εμπλακεί αποφασιστικά στη κρίση της Συρίας η ευρωπαϊκή ένωση όταν η εξωτερική πολιτική της είναι ταυτισμένη με εκείνη των ηνωμένων πολιτειών; Πώς είναι δυνατόν να διατηρηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής όταν όλες τι χώρες της Ευρώπης και κυρίως στην ελλάδα την έχουν κατακλείσει εκατομμύρια μουσουλμάνοι οι οποίοι με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα διακηρύσουν ότι θα επιβάλλουν τον ισλαμικό νόμο της Σαρία σε όλη την ευρώπη πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων όταν ο ίδιος ο κύριος Γιούγκερ είπε ότι πρέπει να έρθουν από τις τρίτες χώρες ε, ταλαντούχοι νέοι. τέλος πώς είναι δυνατόν ο κύριος Γιούγκερ να είναι περήφανος για τη frontex δεν έχει πληροφορηθεί από την ιταλική κυρίως την ελληνική ακτοφυλακή ότι το μόνο που μπορεί να κάνει η frontex είναι να παριστάνει τον τροχονόμο όσων θέλουν να εισέλθουν παράνομα στις δύο αυτές χώρες. ναι πρέπει να γίνει αλλαγή στην ευρώπη αλλά να γίνει με βάση και, ως με κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λαών της και όχι των αιμονών και, και της ιδεολειψίας του ηγετικού κύκλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η διαδικασία Catch the Eye. Και τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει ο πρόεδρος Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα αυτά τα θετικά που είπατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας διαβεβαιώσω τα αρνητικά δεν τα γνώρισα αλλά για λόγους καθαρά περισμού χρόνου δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα. Πάντως από ό,τι συνεπέρανα οι περισσότεροι ευρωβουλευτές εγκρίνουν ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτρέψτε μόνο να πω κάτι για την Τουρκία, γιατί ε, ξέρετε το θέμα της Τουρκίας δεν το έθιξα στην ομιλία μου. Όσον αφορά λοιπόν την Τουρκία, εξακολουθούμε να διεξάγουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά την απελευθέρωση θεωρήσεων. Και θέλω να πω ότι η απελευθέρωση θεωρήσεων θα λάβει χώρα μόνο εφόσον θα έχουν εκπληρωθεί όλες οι ήδη ε, αναφερθήσεις προϋποθέσεις από την Τουρκία. Σε κάποια σημεία βέβαια θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη υπομονή γιατί Πράγματι υπάρχουν δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Τουρκία. Ευελπιστώ ότι θα λυθούν κάπως αυτά τα θέματα, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί. Όσον αφορά, ας πούμε, παραδείγματο χάρη, τη μεταρρύθμιση τη αντιτρομοκρατική νομοθεσία, δεν είναι εύκολο να γίνει μέσα στο προβλεφθέν χρονικό διάστημα και γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι και εύκολο να ορίσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την απελευθέρωση θεωρήσεων όσον αφορά στην Τουρκία. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι σχεδόν όλοι σας επιθυμείτε ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και γνωρίζετε ότι οι διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι ακρογωνιαίος λίθος ε, στην πολιτική μας. Θα περιμένουμε το πέρας των διαπραγματεύσεων και μετά θα καταθέσουμε τις ε, δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ για αυτά που επισημάνατε σχετικά με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Προτείνατε να διπλασιαστούν ή αν θέλετε το προτείναμε εμείς και εσείς συμφωνήσατε ανεπιφύλακτα. Άρα δηλαδή και το Κοινοβούλιο και εμείς οφείλουμε να πράξουμε τα απαραίτητα για να ε, επιτύχουμε το στόχο μας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με το ψηφιακό θεματολόγιο και στο θέμα αυτό οφείλουμε χέρι-χέρι να προχωρήσουμε και να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Πρόεδρε για τη συζήτηση. Πρόεδρος, ε, περνάμε τώρα στον τελικό γύρο ε, της συζήτησης και ξεκινάμε καταρχήν με τους μεγεγραμμένους. Ο κύριος Ζαριανόπουλος παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Χειρότερη η κατάσταση της Ένωσης ομολογήσατε κύριε Γιούγκερ. Ο δικός σας ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ανεργία, φτώχεια, φοροελελασία, ξεριζωμός των αγροτών, τα διέξοδα των νέων με απλήρωτη εργασία και μετανάστευση σίγουρα θα γεροτερέψουν κι άλλο. Και στην Ελλάδα των μνημονίων και παντού. Η Ένωση δεν κινδυνεύει είπατε. Κινδυνεύουν όμως οι λαοί θύματα ανταγωνισμού μεγαθυρίων για ενέργεια και αγορές. Δίνεται μάλιστα κοινό στρατηγείο για επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τους νέους σαν μισθοφόρους εθελοντές για τα θύματά σας τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους στην Ελλάδα. Προτείνεται περισσότερη εκμετάλλευση, φθηνότερου εργαζόμενου, περισσότερα κονδύλια και κέρδη για τα μεγαθύρια, όπω ζητάνε άλλωστε με περισσότερη ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητα παλιά και νέα σοσιαλδημοκρατία ο Λαν Ρέτσι, τώρα και τσίπρας για ενίσχυση των μεγαθυρίων όχι για αυξήσεις μισθών και συντάξεις αφού και αυτοί τσακίζουν τους λαούς τους εξίσου με τη μέρκελ το σόιμπλε και την μέη του brexit. το όραμα όλων σας είναι ο εφιάλτης των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται. Ο καπιταλισμός μόνο ανεργεί, φτώχεια και πολέμους εγγυάται. Η σαπίλα δεν γιατρεύεται, ανατρέπεται. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τα καταφέρει. Έχει εκθέσει τους πολίτες στον τρόμο του Ισλάμ, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που δεν σέβονται ε, τις παραδόσεις μας, νεοναζί στην Ουκρανία, ε, δικτατορία στο Ιράν, ε, αντισημιτική Παλαιστινιακή αρχή, ο Σουλτάνος στην Άγκυρα και από την άλλη μεριά στην Ευρώπη έχουμε χιλιάδες νέους στην ανεργία και πρέπει να πληρώσουμε το λογαριασμό οι Ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο. Ο κύριος Γιούνκερ πρέπει να παραιτηθεί. Αν δεν το κάνει, του ζητώ τουλάχιστον να κάνει τα εξή. Να μην απελευθερώσει τι θεωρήσει για την Τουρκία, την Ουκρανία ή ε, άλλε αλητήριε χώρε. Ε, θα πρέπει να, να στείλουμε πίσω τους ε, μετανάστες ε, και να ενισχύσουμε τα σύνορά μας. Θα πρέπει να πολεμήσουμε τη Ισλαμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λόγο ο κύριο Λέγαμε στην ε, ε, εκστρατεία των Brexit ότι δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό στρατός κλπ. Να, κοιτάξτε το. Ε, ήρθε και αυτό. Ε, το πιο ενδιαφέρον ήταν όταν ο κύριος Γιούνκερ μίλησε για παράλληλες ε, δομές, αλλά το πιο ενδιαφέρον ακόμα ήταν του κύριου Φερχόφστετ που είπε να φύγει η Αμερική, μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας όλα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε παράλληλες δομές χωρίς ανταγωνισμό. Και όταν αποκτήσουμε ανεξάρτητη στρατιωτική αρχή, τότε ε, θα, θα, γίνουμε ισχυροί και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Θυμάμαι, κύριε Φερχόφστατ, ε, ότι με τη Λιβύη θέλατε να σπρώξετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί. Ε, όμως χρειάζεται να στηρίξουμε την ειρήνη και τη συμφιλίωση, όχι αυτά που προτείνονται σήμερα. Μήπως αν κάναμε ε, δημοψηφίσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λαοί θα τα δεχόντουσαν αυτά. Δεν νομίζω. Εκ μέρου των Πρασίνων, το λόγο έχει η κυρία Χάρμ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω κάτι για την Τουρκία. Ξέρετε, αυτή την εποχή μιλάω σχεδόν καθημερινά με συναντέλφου από την Τουρκία αλλά και από την Ουκρανία και νομίζω ότι υπάρχει ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι δημοκρατικέ εξελίξει χώρες όπως είναι η Τουρκία δεν μπορούν να επιβληθούν απ' έξω. Όμως και εμείς έχουμε κάποιες ευθύνες έναντι των δημοκρατών σε αυτές τις χώρες. Έχουμε την υποχρέωση να τους στηρίξουμε και στην Ουκρανία και στην Τουρκία. Ε, δεν μπορούμε να απεκδιώμεθα αυτών των ευθυνών μας. Και κύριε Φαράζ, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Μας λέτε ότι είμαστε εθνικιστές. Ε, να σας πω κάτι, ότι ε, όταν ελήφθη η απόφαση από τους να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά λυπήθηκα. Ε, λυπήθηκα γιατί εσεί ήσασταν εκείνο ε, που υποσχετήκατε στου ε, Βρετανούς ότι τι προκλήσεις του μέλλοντο μπορεί κανεί να τι αντιμετωπίσει με πολιτικέ του παρελθόντο. Και θέλω να σα πω ότι αυτός ο δρόμο, το να γυρίζει κανεί στο παρελθόν ποτέ δεν απέδωσε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής της Υπήρου είναι για εκείνους που θα τολμήσουν γιατί το καλύτερο μέλλον σε αυτή την Ήπειρο ξεκίνησε όταν όλοι από κοινού επιληφθήκαμε ενός κοινού εγχειρήματος. Και λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι αναγκασμένη εγώ Γερμανίδα να το λέω αυτό σε έναν Εγγλέζο ή Βρετανό, αν θέλετε, εθνικιστή. Το λόγο λοιπόν τώρα εκ μέρου ε, τη έχει η κυρία Τσίμα. Δύο παρατηρήσεις θα μου επιτρέψετε. Εγώ ε, δεν νομίζω ότι οι πολίτες ε, θα αισθάνονται καλύτερα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ως ένα είδος δυνατού μειώδους άνδρα ή μορφώματος αν θέλετε. Πάω σε κάτι άλλο, στο PNR. Μιλήσατε εσείς ε, για το ότι είναι απαραίτητο να προστατεύει κανείς ε, την ιδιωτική σφαίρα των ανθρώπων. Ποια είναι η θέση δική σας ε, το ότι η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά σε σχέση με το PNR αντιβαίνει στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει με τον Καναδά. Εκ μέρου των φιλελευθέρων το λόγο έχει ο κ. Φερχόφστατ. Θα είμαι πάρα, πολύ σύντομος. Σοκαρίστηκε η Ρεμπέκα Χάρμς από τα λεγόμενα του κυρίου Φάρατζ. Εγώ όχι. Είναι σαν ε, αλκοολικός ο κύριος Φάρατζ που ε, καταγγέλει κάποιον γιατί πίνει μία μπύρα σε μία pub. Ε, Είπε ο στον πετεινό κεφάλα, όπως λέμε στα ελληνικά. Είναι γελίο. Η πραγματικότητα είναι ότι για τους εθνικιστές και τους λαϊκιστές το θέμα δεν είναι το Brexit, δεν ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα ε, του Βρετανικού λαού και της βιομηχανίας. Ο στόχος είναι να καταστρέψουν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Και αυτόν ε, το στόχο συνεχίζουν να επιδιώκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μας λέει ότι πρέπει να επομιστούμε τις ευθύνες μας ε, για τη γυραιά Ήπειρο και δεν πρέπει να περιμένουμε πάντα από τον Αμερικανικό στρατό να τα κάνει. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνουμε για τη Λιβύη. Ε, για την επιχείρηση. Φυσικά ήσασταν ο καλύτερος φίλος όλων των δικτάτων ανά τον κόσμο και του κύριου Πούτιν. Κύριε Φεχόφστατ, ο κύριος ε, Κάβαλ, Κάβα θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Συμφωνείτε. Κάρβα, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Κάρβα, ε, θέλετε παρακαλώ να δεχτείτε την ερώτησή του. Κάρβερ, ευχαριστώ. Κύριε Φερχόστατες, Συγγνώμη, επειδή θέλετε στενή στρατιωτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σα ενοχλεί ότι έχουμε αυτή την παράδοση τη ουδετερότητα στην Ευρώπη. Για δείτε ε, τι έγινε με τη δημοκρατία τη Ιρλανδία. Ε, ξέρετε τι σημαίνει ουδετερότητα για αυτέ τι χώρε. Ευχαριστώ. Φερχώστατε. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και το ΝΑΤΟ. Εγώ αντίθετα θεωρώ ότι αναπτύσσεται ένα ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ. Είναι απαραίτητο ούτω ώστε να ανακτήσουμε, να ανακτήσουμε τον έλεγχο ε, στην άμεση, ε, στο άμεσο περιβάλλον, στις άμεσα γειτονικές χώρες. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε και όσοι από εσάς ε, συζητάτε στους ε, διαδρόμους ανάμεσα στις ε, θέσεις σας, παρακαλώ είτε να βγείτε έξω είτε να καθίσετε. Εκ μέρου του ECR το λόγο έχει ο κύριος Καμάλ. Χαίρομαι που μιλώ μετά τον κύριο Φερχόφστατ. Μια και ξεπεράσαμε την ομάδα του Ευρωπαϊκής Κοινοβούλια στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου σε ψήφους. Ε, αν συνεχίσετε να αναγνωρείτε τις ανησυχίες του κόσμου, αν συνεχίσετε να ε, προωθείτε την ολοκλήρωση αντί να δημιουργείτε θέσεις εργασία, τότε πράγματι οι ψηφοφόροι θα πέσουν στα χέρια αυτών που ονομάζεται λαϊκιστές. Ναι, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό όμως ε, δεν είναι ουδέτερο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ε, και οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Βασίλειο χρειάζονται πολιτικέ για την απασχόληση, για την ασφάλεια, για νέες ευκαιρίες. Αυτό προ όφελο όλων των χωρών που βρίσκονται, αντιπροσωπεύονται εδώ σήμερα. Φοβάμαι όμω ότι σήμερα ακούσαμε πάλι τα ίδια λόγια. που ακούμε πάντα εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριο Πιτέλα. Ε, πραγματικά μένω ενεό ακούγοντας κύριε Πρόεδρε τον συνάδελφο κύριο Φάρατζ και τη συνάδελφο κυρία Λεπέν να ισχυρίζονται βοηθήστε μας, βοηθήστε μας ε, για να υλοποιήσουμε το Brexit. Μα λυπάμαι πάρα πολύ, αυτοί ήταν οι αποφασισμένοι, οι αμετακίνητοι στο να ζητούν η μεν το Brexit και η κυρία Λεπέν το Frexit και τώρα λένε ότι δεν τα καταφέρνουν ε, και ε, θέλουν να έχουν συμμαχία με τον διάβολο, με τον κύριο Φερχόφτσετ, μα εσείς είστε ο διάβολος, εσείς μας εξαπατήσατε εξαπατήσατε και εξαπατήσατε και τους Βρετανούς με τα ψέματά σας και τους οδηγήσατε σε μια κατάσταση που θα είναι ζημιά και για τους Βρετανούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο έχει σχέση με τη φτώχεια, με την κατανομή του εισοδήματος, το κοινωνικό τάμπινγκ, την ανάπτυξη, ε, τη βιοφόρα ανάπτυξη. Αυτά είναι δικέ μα προτεραιότητες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιούγκερ γιατί αυτά είναι προτεραιότητες και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτο τώρα. Σήμερα το πρωί εισαγάγατε την ε, Capital Market Union όπως την αποκαλέσατε. Ε, τώρα έχουμε να ολοκληρώσουμε πρώτα ε, την κοινή αγορά, μετά την κέφαλη αγορά. Ε, θα πρέπει ε, βέβαια, εντάξει αυτά, αλλά να δουλέψουμε για την πολιτική ένωση, την ενοποίηση, την πολιτική. Ίσως πείτε ότι ο κ. Πιτέλα ονειρεύεται. Ναι, ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, για καλύτερα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δύναμη εκείνη που θα μας επιτρέψει να παραμείνουμε ενωμένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όπως έλεγε ο Ντελόρ, χέρι-χέρι, αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταγάγουμε νίκη και μπορούμε ακόμα να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Πρόεδρος, το λόγο έχει για το ΕΛΚ ο κύριος Βίμπα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, ε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, εμένα αυτό που μου άρεσε σήμερα στη συζήτηση ήταν ε, αυτό το σοβαρό ύφο. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι περιμένουν να του δώσουμε απαντήσει. Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι ο κύριο Γιούγκερ με το πρόγραμμά του, ε, με την υποστήριξη αυτού του Κοινοβουλίου και με τη βοήθεια των υπολείπων μπορεί να ξεκινήσει την πραγματική δουλειά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε οι δυο μα, οι δύο θεσμοί. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό μετά από μια συζήτηση τριών ετών. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να δούμε κατά πόσον και τα κράτη-μέλη θα κινητοποιηθούν. Αυτή η συζήτηση που γίνεται βορρά-νότου για την Ευρωζώνη, Ανατολή-Δύση για το προσφυγικό και πριν από λίγε μέρε κάποιο σκέφτηκε και όλο να ζητήσει την εκδίωξη ενό κράτου-μέλου. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά μερικέ φορέ έχω την ότι δεν είμαστε σε νηπιαγωγείο και δεν είμαστε σοβαροί πολιτικοί. Γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο επιτέλου πρέπει να βρει τι κατάλληλε απαντήσει τα σημεία των καιρών. Ε, και κυρίε και κύριοι, όσον αφορά την αντιπαράθεσή μα με του λαϊκιστέ και του ακραίου αριστερά και δεξιά, θέλω καταρχήν να σας πω ότι όσον αφορά στο Brexit, ε, να μην μου θυμώνετε, αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με εκείνου που λένε ότι οι επιπτώσεις στο σύνολο της Ευρώπης θα είναι, με βάση τις δημοσκοπήσεις που έγιναν σήμερα, θα είναι λοιπόν οι επιπτώσει αυτές που δείχνουν ότι οι περισσότεροι το εγκρίνουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ε, στη δική μου τη χώρα από το 77 δεν είχαν πει τόσοι πολλοί άνθρωποι ότι δεν τους νοιάζει καθόλου. Και ξέρετε γιατί, διότι οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη βλέπουν ότι το πρόβλημα δεν θα είναι του Βερολίνου, ούτε και του Παρισιού, αλλά ούτε και της Ρώμης. Οι πολίτες βλέπουν ότι το Λονδίνο θα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή το πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφωνίες, τσακωμοί στο Λονδίνο, ακόμα και οι πρωταγωνιστές της εξόδου, ε, ε, τα σημαντικότερα μέλη αποσύρονται. Ο Φαράτς αποσύρεται. Τζόνσον ούτε τον ακούμε. Ο κύριο Φαράτσου λέει, ξέρετε αυτά τα 460 εκατομμύρια που δίθεν τα εξοικονομούσαμε, αυτό σα το είπα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη συζήτηση για τον Brexit θα την μετωπίσουμε θετικά. Αν μια χώρα θέλει να φύγει, ε, τότε να μην λένε μόνο οι Βρετανοί Brexit σημαίνει Brexit, να του λέμε και εμεί Brexit, ξέρετε Brexit, αφήγετε. Και αυτό θα είναι δύσκολο για εσά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που θα πρέπει να απαντήσει στο μέλλον ο κύριο Φάρατζ στα παιδιά του. Να του εξηγήσει τι ακριβώς επέφερε στην πατρίδα του. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι όπως τα έκανε και ο κύριος Γιούγκερ πρέπει να διατηρήσουμε τις αρχές μας. Εμείς στηρίζουμε την Ευρώπη και η συζήτηση για τον Brexit θα καταδείξει ότι είναι σωστή και η συζήτηση που γίνεται για την Ευρώπη. Κύριε Βίμπα ο κύριος Κόμπορν ε, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση, γιατί είναι ένας από αυτούς, ε, επειδή είναι ένας από αυτούς που κάποτε θα φύγουν, σας παρακαλώ, δεχτείτε την ερώτησή του. Παρακαλώ κύριε Κόμπουνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Herr President. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί τελευταία το Παρίσι. Εγώ έχω να πάω αρκετό καιρό. Αλλά κυκλοφορώντα το Παρίσι, αλλάζοντα τρένα, με εξέπληξε ο αριθμό των ανθρώπων που κοιμούνται έξω στο δρόμο αυτό δεν είναι πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τους νέους, οι νέοι στηρίζουν τον Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλο και περισσότεροι στη Γαλλία και σε άλλες χώρες κάνουν το ίδιο. Δεν συμφωνείτε μαζί μου. Ο κύριος Βίμπα έχει το λόγο. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι κανονικά δεν αξίζει καν τον κόπο το να δίνει κανείς ε, στους λαϊκιστές ε, χρόνο για να ρωτάνε στο πλαίσιο μιας μπλε Ίσως πρέπει να το σκεφτούμε αυτό στο μέλλον. Παρόλα αυτά, Μισό λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος διακόπτει. Ε, ο κύριος Βίμπα, βεβαίως, ε, βλέπετε πώς δουλεύουν οι λαϊκιστές και οι εξτρεμιστές. Στρεβλώνουν την πραγματικότητα, προβαίνουν σε απλουστεύσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα κόσμο που είναι περίπλοκος και γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο που έχουμε χαράξει. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Κύριε Βίμπα, σε αυτή την αίθουσα ε, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί μια ερώτηση. Είχατε το δικαίωμα να πείτε όχι, δεν μου κάνει κέφι, δεν έχω καμία όρεξη να απαντήσω στην ερώτηση. Αλλά ε, οι συνάδελφοι θα πρέπει να το σκεφτούν ότι τίθενται κάποιες ερωτήσεις ακόμα και αν δεν αρέσουν. Πολύ ωραία λοιπόν.